Άρχεται η συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας. Σας καλωσορίζω θερμά αγαπητοί συνάδελφοι. Και ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η αυριανή συνεδρίαση της 5ης 4 Δεκεμβρίου ακυρώνεται εξαιτία ε, διαγραφή κάποιων σημείων από την σε διάταξη. Το σημείο 12, ε, συνάντηση με την ε, Ιταλική Γερουσία και Βουλή, γιατί οι προσκυκλημένοι μας είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις, οπότε δεν μπορούν να έρθουν αύριο. Ακυρώνεται αυτό το σημείο και άρα αναβάλλεται η αυριανή σε διάταξη. Επίσης, τα σημεία 13 και 14 οι νομοθετικές προτάσεις για την κλωνοποίηση. Λόγω της απόφασης της διάσκεψης των Προέδρων για την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 55 για την κοινή συνεδρίαση επιτροπών περιβάλλοντος και γεωργίας. Εξαιτής λοιπόν αυτών των αλλαγών χρειάστηκε να κυρώσουμε την αυριανή μα συνεδρίαση. Περάμε στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης, την έγκριση των πρακτικών της 6ης και 7ης Οκτωβρίου. Ως ήθιστε, αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις για τα πρακτικά, θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα. Έχουμε αναμετάδοση από το διαδίκτυο της συνεδρίασής μας και εξασφαλίζεται διερμηνία σε 19 γλώσσες με εξαίρεση δεστονικά, λετονικά, μαλτέζικα και σλοβακικά. Σημείο 4. Αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις για τη δημοκρατία της Μολδαβίας. Ο κύριος Ρεμπέγκα είναι εισηγητής της γνωμοδότησης αυτής. Θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Μετά την ψηφοφορία θα επιδώσουμε την γνωμοδότησή μας στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου που είναι αρμόδια επί της ουσίας ε, και θα συζητήσει αυτό το θέμα αυτή τη βδομάδα. Δεν ξέρω αν ο εισηγητής μας ο κύριος Ρεμπέγκα έχει κάποια σχόλια. Αν έχει κάτι να προσθέσει, έχει το λόγο ή δεν μη. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Αλλά μια στιγμή ο κύριος Φεράν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με τον συνάδελφό μου έχουμε υποβάλει μια τροπολογία και θα ήθελα απλώς να παρουσιάσω την τροπολογία, ούτως ώστε όλοι να γνωρίζουν ποιο είναι το έτοιμά μας. Θέλουμε να επενθυμίσουμε ότι οι ενισχύσει που έχουμε απελευθερώσει για τους Ευρωπαίους Γεωργούς όσον αφορά το πάρκο της Ρωσίας ε, και τιμή των τιμών ήταν επαρκές. Θέλουμε να θαρρύνουμε τις αγωγές από τη Μολδαβία, να μειώσουμε τους τελωνιακούς δασμούς και αυτό ίσως οδηγήσει ε, σε μια επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τους Ευρωπαίους γεωργούς και εμείς καλούμε να υπάρξει υποστήριξη των Ευρωπαίων αγροτών. Σας ευχαριστούμε κύριε Φερά. Μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα. Ψηφίζουμε λοιπόν την ε, γνωμοδότηση αυτή για τις αυτόνομες προτιμήσεις, ε, εμπορικές προτιμήσεις ε, για τη διαδικασία της Μολδαβίας. Ο κύριος Μπονάνο ζήτησε το λόγο. Συγγνώμη που δεν ζήτησα το λόγο προηγουμένω. Εγώ συμφωνώ απόλυτο με εκείνο που είπε ο συνάδελφος κ. Φεράν όσον αφορά την ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει δυσκολίες και το ρωσικό εμπάργκο είναι μεγάλη ανοησία. Τελικά την πληρώνουν μόνο οι Ευρωπαίοι ε, αγρότες. Ε, και στο τέλος ε, το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει με το ρίσκο και την πληρώνει ο κόσμος. Λοιπόν, θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ε, που αφορά την υγεία και εγώ και είμαι δήμαρχος. Όλοι θα εξηγήσουν ε, τις ε, διακόπτη κάποιους, όλοι θα εξηγήσουν τις τροπολογίες. Δεν θα, δεν θα τελειώνουμε ποτέ να εξηγούμε τις τροπολογίες κύριε Πρόεδρε, να ψηφίσουμε. Μπορώ να μιλήσω ή όχι. όχι, σταματήστε, μην μιλάτε. Μα ποιος μιλάει. Εδώ τα ταμπέλα φίλος. Ε, όπως συνήθως μας τις πάει. Εσύ μας τις πας. Σκάσε, εσύ μας τις πας. Εσύ και οι φίλοι σου μας τις πάτε. Μπορώ να να, τελειώσω, να μιλήσω. Παρακαλώ, ησυχία παρακαλώ. Σας έδωσα το λόγο γιατί νόμιζα... Νόμιζα ότι ήταν ένα διαδικαστικό θέμα. Δεν θα αρχίσουμε τώρα συζήτηση επί της ουσίας, παρακαλώ. Συζήτηση επί της ουσίας δεν επιτρέπεται τώρα. Νόμιζα ότι θέλατε το λόγο για ένα διαδικαστικό θέμα και συγγνώμη, έκανα λάθος. Γνωρίζουμε όλοι τους κανόνες, αυτό θεωρούσα τουλάχιστον. Κάποιο ζήτησε το λόγο, ακριβασκόπημα να του το δώσω. Αλλά όχι τώρα για να ξεκινήσουμε συζήτηση επί της ουσίας. Αρκούσε μία παρατήρηση, δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε όλη τη συζήτηση. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία, ψηφίζουμε την πρώτη τροπολογία. Ποιος είναι? Να μιλήσω κάτι διαδικαστικό, παρακαλώ. Επιτρέπετε. Θα ήθελα να ολοκληρώσω κάτι. Eh, ακουστικά που είναι εδώ, καθαρίστε τα. Διότι είναι απέσιες, ε, από, πρέπει κάποιο να τις καθαρίσει, είναι κακό για την υγεία και εδώ και στο Στρασβούργο και στην Ολομέλεια. Είναι βρώμικα τα ακουστικά. Μετά μιλάτε για καθαριότητα. Άλλη μια νοητεία. Θα ψηφίσουμε, πάψε. Εδώ είμαστε για να μιλάμε, όχι για να φλιαρούμε. Πάρε ένα βάλιουμ να ηρεμήσει, ραμπελα, Πάρε βάλιουμ. Είναι πρωί. Δεν είναι σημαντικό. Δεν... Είναι κρίμα να αρχίζουμε να χωνόμαστε από τόσο νωρίς το πρωί. Παρακαλώ, Σα επαναφέρω στην τάξη. Α δείξουμε όλοι μια ευπρεπή συμπεριφορά. Ποιο είναι υπέρ της πρώτης τροπολογία, ποιο είναι υπέρ. Διανατάσσεω της χειρό, Κατά. Κατά. Αποχές από την πρώτη τροπολογία. Απορρίπτεται η πρώτη τροπολογία. Περνάμε στη δεύτερη τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, ευχαριστώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ, κατά, Απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 4. Ποιος είναι... Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. τελική ψηφοφορία του σχεδίου γνωμοδότησης ε, με τις τροπολογίες. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Αν δεν έχει κάποιος την κάρτα του, να το δηλώσει για να συμπεριλάβουμε την ψήφο του. Αν έχετε τις κάρτες σας, παρακαλώ, ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ, έχουμε ψήφους που περισσεύουν. Ε, κάποιος από το ΕΛ και κάποιος από τους σοσιαλιστές παρακαλώ να μην ψηφίσει. Εντάξει τώρα. 35 ψήφισαν υπέρ, 5 κατά και 2 αποχές. Σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση του κυρίου Ρεμπέγκα. Και παρακαλώ, θέλουμε και στο μέλλον να τηρήσουμε και να τηρούμε τους κανόνες, γιατί υψηλή τόνη και η αγένεια δεν είναι σωστό να επικρατούν στην Επιτροπή μας. Περνάμε στο επόμενο σημείο, σημείο 5, δημόσια ακρόαση για τα βιολογικά προϊόντα και την σήμαση, την ετικετοθεσία των βιολογικών προϊόντων. Με ιδιαίτερα χαρά θα κηρύξω την έναρξη της δημόσιας ακρόασής μας για τη νέα πρόταση του κανονισμού για την βιολογική παραγωγή και τη σήμανση των βιολογικών προϊόντων. Οργανώνουμε αυτή την δημόσια κρόση στα πλαίσια της προετοιμασίας μας, της νομοθετικής μας έκθεσης, για την οποία αρμόδιος συγητής είναι ο κύριος Χόισλινγκ. Μια στιγμή γιατί δεν χωράνε όλοι οι καλεσμένοι μας δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις όρθιοι θα μπορούσαν ίσως να καθίσουν ε, όπου βρουν και νέες θέσεις για να μην έχουμε ορθίους στην αίθουσα. Παρακαλώ γραμματεία να περιποιηθεί τους καλεσμένους για να μην μένουν όρθιοι. Έχουμε και την κυρία Πιετικάινεν που είναι η συντάκτηρη της γνωμοδότησης Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος και έχουμε και την κυρία Μάη στη συνεδρίαση που είναι η συντάκτηρη της γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών. Έχετε λάβει το πρόγραμμα της ακρόασης. Θα ήθελα να καλωσορίσω ολόθερμα τους εμπειρογνώμονές μας, τους οποίους εντός ολίγου θα ακούσουμε για τις παρουσιάσεις. Θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Χόισλινγκ όπως είπα, και στη συνέχεια θα ακούσουμε την συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής ΕΜΒΗ, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, την κυρία Πιετικάινεν και ακολούθως την κυρία Μάη, την συντάκτρια γνωμοδότηση από την Επιτροπή των Περιφερειών. Πρώτα όμως, ο λόγος στον κύριο Χόισλινγκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο και ευχαριστώ πολύ για τον ενδιαφέρον που έχετε δείξει για αυτήν εδώ την ακρόαση. Βλέπω η αίθουσα είναι γεμάτη και έχει να κάνει λοιπόν η ακρόαση με την πρόταση φέτος την άνοιξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αλλαγή του κανονισμού για τα βιολογικά προϊόντα. Αυτή η πρόταση έχει οδηγήσει σε πάρα πολλές συζητήσεις και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμούμε να αλλάξουμε την πρόταση κανονισμού αυτή με πρακτικές τροποποίησεις. Η συζήτηση λοιπόν ήταν πάρα πολύ έντονη για τα βιολογικά προϊόντα, ιδιαίτερα για τις οριακές τιμές που χαρακτηρίζουν τα βιολογικά προϊόντα. Εμείς θέλουμε μηδενικές τιμές. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθούν όλοι οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα προϊόν βιολογικό. Οι οριακές τιμές λοιπόν είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό που έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλες συζητήσεις. Και μεταξύ αυτών της στη σημερινή ακρόαση. Χρειάζεται ένα σαφέστερος ορισμός αυτών των οριακών τιμών και σε αυτή την ακρόαση θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις. Επίσης, οι, τα οι τροφές οι ζωοτροφές είναι θέμα αυτής της ακρόασης. Και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης θα ασχοληθούμε με το θέμα των πράξεων κατεξουσιοδότηση, οι οποίες είναι αρκετά προβληματικές. Πάντα σε σχέση με τον κανονισμό για τα βιολογικά προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει κάποιες ε, πολύ γενικές ε, διατάξεις για τον κανονισμό και εμείς θέλουμε να προσπαθήσουμε να τις αναλύσουμε και τις περιορίσουμε. Επίσης, το θέμα του ελέγχου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο έλεγχος των βιολογικών προϊόντων αποτελεί αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη προς το παρόν και είναι κάτι που έχει προκαλέσει μεγάλες ανησυχίες, διότι ο έλεγχος για τα βιολογικά προϊόντα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του κανονισμού Χρειάζεται βελτίωση, σε αυτό συμφωνούμε όλοι, όμως πιστεύω πως ε, είναι λάθος να μεταφερθεί αρμοδιότητα σε άλλες ε, γενικές ε, διευθύνσεις. Στην Ευρώπη η βιολογική γεωργία είναι μία βιομηχανία η οποία ολοένα και μεγαλώνει. Αυτό φυσικά είναι καλό αλλά δημιουργεί και πάρα πολλές προκλήσεις και ο κανονισμός πρέπει να έχει ως σκοπό να πλουστεύσει την κατάσταση και όχι να τη δυσκολέψει. Πιστεύω ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ήδη αναλάβει δράση και έχουμε ήδη αρχίσει τις συζητήσεις. Το Συμβούλιο μας ακολουθεί. Πρέπει να ακούσουμε τις ανάγκες και των παραγωγών αλλά και των καταναλωτών και πιστεύω πως ε, όταν συνδυαστούν αυτές οι ανάγκες θα καταφέρουμε να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα για το πώς, για το πώς πρέπει να είναι αυτός ο κανονισμός. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. είναι ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο και για την κοινωνία και γι' αυτό είναι σημαντικές οι παρατηρήσεις του εισηγητού γιατί οι συμπολίτες μας ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Πιετικάιν τη συντάκτρια γνωμοδότης από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Καλώς ήρθατε κυρία Πιετικάινεν. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτή την κοινή ακρόαση και προσβλέπω σε πολύ στενή συνεργασία με την Επιτροπή Γεωργίας επί του ζητήματος. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι βιολογικές αγορές αυξάνονται ταχαίως στην Ευρώπη και πράγματι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό μπορεί να συνεπιφέρει πρόσθετο εισόδημα στους ε, παραγωγούς και τους γεωργούς που παράγουν βιολογικά προϊόντα και στο μέλλον επίσης μπορεί να είναι ο δρόμος για τις εξαγωγές ε, της παραγωγής τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων της ε, Ευρώπης σημαίνει αύξηση όσον αφορά τη ζήτηση των καταναλωτών και θα αυξάνεται και το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα καλά τρόφιμα, τρόφιμα για τα οποία γνωρίζουν την προέλευσή τους, τα βιολογικά προϊόντα. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η ποιότητα των βιολογικών τροφίμων είναι καλή και για μένα ένα από τα σημαντικά στοιχεία είναι πώς θα ασχοληθούμε με τους ελέγχους και τις ε, απάτες. Ε, όλοι γνωρίζουμε ότι όλοι οι γεωργοί και οι παραγωγοί στην Ευρώπη κάνουν ό,τι μπορούν. Δεν πρέπει να τους ε, αυξήσουμε το άχθος με λεπτομερείς ελέγχους και αύξηση των ελέγχων. Η προσέγγιση που εισάγεται εδώ με βάση τον κίνδυνο είναι πάρα πολύ καλή. Θα πρέπει να είναι αυστηρότερη όμως η έλεγχη, κυρίως όσον αφορά τα προϊόντα από εισαγωγές από τρίτες χώρες θα θυμόσαστε το σκάνδαλο με το κρέας αλόγων. Ε, εάν υπάρξει κάποιο σκάνδαλο, ε, βλάπτει επί μακρό χρονικό διάστημα όλη την παραγωγή. Καταλαβαίνω σαφώς ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αμέσως εδώ τις αλλαγές εντός αυτού του κανονισμού. Ελπίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να ελπίσουμε θα κάνουμε τα επόμενα βήματα. Να έχουμε μια κοινή πολιτική τοποθέτηση. Να αναπτύξουμε εσωτερικές, εσωτερικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα. Τι σημαίνει αυτό. Τι ούτω τρόπος μπορούμε να πετήσουμε αυστηρότερους ελέγχους από τις περιοχές εκείνες που είναι εκτός του κανονισμού που δεν μπορούν να είμαστε βέβαιοι για την προέλευση των προϊόντων. Οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν εσωτερικό σύστημα ελέγχου και επιθεωρήσεων. Και αυτό θα πρέπει να ελέγχεται από το τρίτο μέρος και θα επιβάλλονται κυρώσει στο τρίτο μέρος που διενεργεί τους ελέγχους και που θα πρέπει να είναι ε, εγγεγραμμένος ο φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταχωρημένος. Αυτό είναι θέμα ε, που κάνουμε και σε άλλους οικονομικούς τομείς. Κάνουν, έχουμε τον εξωτερικό έλεγχο των εταιριών που κάνουν τον εσωτερικό τους ε, λογιστικό έλεγχο και είναι υπεύθυνε οι εταιρείε να ελέγχουν το ισοζύγιο του και το πώς γίνονται εσωτερικοί έλεγχοι. Δεν στέλνουμε συνεχώς εξωτερικούς ελεγχτέ εταιρείε να κάνουν τους ελέγχους. Κάτι παρόμοιο πρέπει να κάνουμε εδώ. Και πρέπει να στείλουμε έτσι, προσεγγίζοντας έτσι το θέμα, το σωστό πολιτικό μήνυμα. Κάποια άλλα σημεία που θα ήθελα να θίξω. Έχουμε κάποιες λεπτομέρειες που θα πρέπει να εξετάσουμε στην κοινοβουλευτική μας εργασία. Ένα θέμα είναι το εξής. Σε όλη την εκμετάλλευση θα πρέπει να έχει βιολογικές καλλιέργειες. Υπάρχει σύστημα που ένα τμήμα της εκμετάλλευσης έχει βιολογική καλλιέργεια και έτσι μπορούμε να διευκολύνουμε την, ε, μετατροπή της εκμετάλλευσης σε μια εκμετάλλευση που θα παράγει μόνο βιολογικά προϊόντα. Αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε λεπτομερέστερα. Μετά είναι οι σπόροι και το αναπαραγωγικό υλικό. Εάν προβλέπονται αυξανόμενες ανάγκες, άρα θα πρέπει να έχουμε επικοιλωμορφία. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε σπόρους και αναπαραγωγικό υλικό που είναι εκτός του βιολογικού φάσματος ενδεχομένως, αλλά θα πρέπει να μετατρέπεται σε βιολογικό το ταχύτερο δυνατόν. Και κάτι άλλο, και την παραγωγή αερίων, την παραγωγή στα θερμοκήπια. Και ποιος κανονισμός θα μπορεί να καλύπτει την βιολογική παραγωγή. Ελπίζω και αυτόν το εξετάσουμε μαζί θα μπορούσαμε κάπου να βελτιώσουμε το κείμενο, να έχουμε σαφέστερους ορισμούς όσον αφορά την ευημερία των ζώων και τι προσδοκίες υπάρχουν. Βιολογικό δεν σημαίνει η χημική συνιστόσα της παραγωγής, αλλά σημαίνει επίσης και το πώς διαμορφώνεται η όλη η αλυσίδα της παραγωγής. Υπάρχουν πολλά θέματα που τίθενται Κάποιες είναι απλώς μικρολεπτομέρειες. Πρέπει να εξετάσουμε κάποιους ορισμούς και να προβούμε σε κάποιες διευκρινήσεις. Δεν θα αναφερθώ τώρα σε λεπτομέρειες. Απλώς ε, όπως και προηγούμενος μιλητής, θέλω να πω ότι το θέμα των κατεξισοδότης συμπράξεων θα πρέπει να εξεταστεί επίσης και να αποφασίσουμε κατά πόσο έχουμε προχωρήσει πολύ μακριά όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και προσβλέπω στα σχόλιά σας και την ακρόαση και στην καλή μας συνεργασία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα λάβει σύντομα το λόγο και η κυρία Μάης, που είναι συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών. Είναι εδώ η κυρία Μάης. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, ευκαιρία που μου δίνετε. Να σας πω δύο λόγια για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Είμαι μέλος της Επιτροπής Περιφερειών και αρμόδια εισηγήτρια για τη... τον κανονισμό αυτό. Αύριο θα εξετάσουμε στην ε, Επιτροπή των Περιφερειών την έκθεσή μου για να δούμε ποια σημεία είναι σημαντικά για μας. Αυτό που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο κανονισμός είναι άμεση εφαρμογής, ε, γι' αυτό και τα αποτελέσματα θα φανούν αμέσως στις περιφέρειες. Συμφωνούμε με την ιδέα, έχουμε κάποιες επικρίσεις για τους συγκεκριμένους τρόπους ε, εφαρμογής. Καταρχήν, το θέμα της παράλληλης γεωργίας. Η Επιτροπή θέλει να σταματήσει αυτή τη δυνατότητα, ενώ σε ορισμένες περιοχές το 40% της παραγωγής ε, είναι μεικτή παραγωγή. Θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στις περιφέρειες αυτές ε, που δεν θα μπορούν πια να επιτρέπουν βιολογική παραγωγή. Δεν μπορούμε να έχουμε 100% ε, βιολογική παραγωγή μέχρι το 2020 όπως ε, ζητά με υπερβολικά φιλόδοξο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε ένα πιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Η, η Επιτροπή των Περιφερειών δεν θέλει ειδικού κανόνες ε, για τα βιολογικά τρόφιμα σε σχέση με άλλα ποιοτικά τρόφιμα. Γιατί αν δημιουργήσουμε διάφορα επίπεδα προστασίας θα προκαλέσουμε σύγχυση στον καταναλωτή. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να θεσπίσει ε, μία υποχρέωση αποτελέσματος ε, επιδόσεων. Δυσεφάρμοστο θα είναι όμως αυτό το θέμα στην πράξη, γιατί οι βιοκαλλιεργητές δεν είναι αποκομμένοι από τον κόσμο και νομίζω ότι είναι άδικο να τους ε, επιβαρύνουμε με οικονομικές ευθύνες που θα τους ξεπεράσουν. Επίσης, θέλουμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία για τους μικροκαλλιεργητές. Συμφωνώ, αλλά ο ορισμός προβλέπει τα 5 εκτάρια καλλιεργήσιμη γη. 5 εκτάρια όμως σε ορισμένες χώρες είναι μεγάλη έκταση. Σε μικρές χώρες για παράδειγμα, ενώ στη Γαλλία 5 εκτάρια είναι μια μικρή καλλιέργεια. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε περισσότερη υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες και τις διαφορές. Καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο αναφοράς το τζίρο, τον κύκλο εργασιών και όχι την ε, αγροτική επιφάνεια. Επίσης, το θέμα του εμπορίου με τις τρίτες χώρες θα πρέπει και στο σημείο αυτό να εξασφαλίσουμε διαφάνεια. Γιατί δεν έχουμε τέτοια διαφάνεια. Το ίδιο προϊόν τη χάνει διαφορετική μεταχείρισης ανάλογα από το που προέρχεται. Θα πρέπει ο καταναλωτής να είναι σίγουρος ότι θα έχουμε ίση μεταχείριση για ισοδύναμα προϊόντα από όπου και αν προέρχονται. Καλό θα ήταν να διατηρήσουμε τους ετήσιους ελέγχους που εφαρμόζουμε σήμερα και να μην χρησιμοποιούμε υπερβολικά τη μέθοδο της αξιολόγησης κινδύνου. Εφτά σημεία ανέφερα, τα πιο προβληματικά κατά τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών σε ό,τι αφορά τον κανονισμό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία με την έκθεση. Αν εγκριθεί ο κανονισμός ως έχει, ίσως δημιουργήσει προβλήματα γιατί θα οδηγήσει στην ε, εξαφάνιση κάποιων προϊόντων από την εσωτερική αγορά και θα μας υποχρεώσει να εισαγάγουμε αυτά τα προϊόντα έξωθεν. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν άδικο για πολλές περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Είναι χρήσιμη η γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, των Περιφερειών γιατί και το δικό σας θεσμικό όργανο ε, επηρεάζει με τη γνώμη του τα θέματα αυτά. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τους εμπειρογνώμονές μας. Πρώτα δύο, θα ακολουθεί η συζήτηση για κατόπιν τους άλλους τρεις. Πρώτα έχουμε τον εκπρόσωπο από τη Γερμανία, τον Γερμανικό Σύνδεσμο Βιολογικής Οικονομίας Τροφίμων. Ο πρώτος μας καλεσμένος είναι ο κύριος Φέλιξ Πρίντσου Λεβενστάιν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε να έρθω εδώ σε αυτή την ακρόαση και να σας παρουσιάσω τη θέση του γερμανικού βιολογικού κλάδου και εν μέρη του ευρωπαϊκού βιολογικού κλάδου τροφίμων. Προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που μας ε, δόθηκαν με τις δικές μας εκτιμήσεις. Πρέπει να πω ότι από τον κανονισμό έχει προκύψει το ερώτημα του εάν η βιολογική γεωργία είναι η εναλλακτική λύση. Και εάν θα έχει την στήριξη που χρειάζεται από καταναλωτές και παραγωγούς οι εξελίξεις στην συμβατική γεωργία ήταν ε, δραματικές και για την ε, βιοπικιλότητα και για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων και για την κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε την βιολογική γεωργία για το καλό όλη, όλου του κλάδου της γεωργίας. Είναι αναγκαίες αυτές οι αλλαγές και αυτό το δείχνουν πάρα πολλές μελέτες, ένα και αυξανόμενος αριθμός μελετών. και υπάρχει ένα ανεκμετάλλευτο δυναμικό στη βιολογική καλλιέργεια, το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης της βιολογικής καλλιέργειας, η οποία, η οποία πρέπει να βγει από αυτόν τον μικρό θύλακα στον οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Φυσικά, χρειάζεται να στηρίξουμε την αξιοπιστία της βιολογικής καλλιέργειας και αυτό σημαίνει να αυξηθεί, να αυξηθεί ο έλεγχος, να αυξηθεί η ποιότητα του ελέγχου και να απαγορευτούν οι μικτές ε, καλλιέργειες, η μεικτή παραγωγή. Σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης υπάρχει απαγόρευση των μεικτών καλλιεργειών και αυτό αυτή είναι μια τάση που όλο ένα και αυξάνεται. Επίσης, η τρίτη ερώτηση που μας ετέθη ήταν για, τα, για τις οριακές τιμές καταλήπων. Για να χαρακτηριστεί βιολογικό ένα προϊόν χρειάζεται ο παραγωγός να παραμείνει εντός των οριακών τιμών καταλήπων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να, να του τους ε, αγρότες υπεύθυνου για αυτές τις τιμέ καταλήπων είναι για μας δικαιολόγητη και θα παρεμποδίσει και νέους ε, αγρότες να ασχοληθούν με τη βιολογική καλλιέργεια. Εμείς, θα σας δώσω ένα παράδειγμα από την δική μας ε, περίπτωση. Εμείς παράγουμε διάφορα χορταρικά και καρικεύματα. Όταν αυτά περιέχουν εθέρια έλαια, για παράδειγμα μέντα, τότε μέσα σε αυτά τα εθέρια έλαια βρίσκονται διάφορα λιποδιαλυτά συστατικά, τα οποία έχουν μεταφερθεί από το περιβάλλον. Και αυτό, αυτή η μεταφορά είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. επίσης, όταν εγώ έχω έναν αγοραστή, ο οποίος θέλει να αγοράσει αυτό το προϊόν, αυτή τη μέντα, τότε, εάν εκείνος βρει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους στο προϊόν ε, το οποίο θα αγοράσει ε, οριακές τιμές υψηλότερες, τότε θα αποσυρθεί όλη η παρτίδα από την αγορά. Και αυτό φυσικά ζημιώνει και τον ε, παραγωγό και τον αγοραστή. Υπάρχει λοιπόν ένας ε, κίνδυνος τόσο στη δειγματοληψία για τον ε, έλεγχο του αν ένα προϊόν είναι βιολογικό πραγματικά και στον ε, έλεγχο των οριακών αυτών ετοιμών. Πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός και να δημιουργηθούν ε, νέοι τρόποι ελέγχου αυτών των οριακών τιμών. Ε, και φυσικά δεν πρέπει αυτές οι οριακές τιμές να χρησιμοποιηθούν για να ασκηθεί πίεση στους παραγωγούς. Πιστεύουμε πως εδώ πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η αρχή του οριπένων πληρώνει. Αλλά οριπένων σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να είναι ο παραγωγός, ο οποίος δεν μπορεί να ελέγχει το περιβάλλον. Διότι υπάρχει και περίπτωση, για παράδειγμα, ενός βιολογικού αμπελουργού, ο οποίος ε, όταν μία χρονιά η παραγωγή του δεν πάει καλά, δεν θα έχει καθόλου ε, προϊόν. Δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να λύσουμε αυτό το πρόβλημα προς το παρόν και δεν υπάρχει δυνατότητα να ε, λυθεί ούτε δικαστικά. Πρέπει να γίνει μια συνολική αναπροσαρμογή αυτού του συστήματος οριακών τιμών. Τώρα, όσον αφορά το σύστημα ελέγχου, φυσικά χρειάζεται ε, αυτό το σύστημα ελέγχου των οριακών τιμών να είναι αυτό ακριβώς, να είναι ένα σύστημα ελέγχου. Υπάρχει αυτός ο δειγματοληπτικός ε, έλεγχος που ισχύει αυτή τη στιγμή και σε γενικές γραμμές, ναι, μπορούμε να πούμε πως είναι ε, πολύ καλό το ότι η βιολογική γεωργία έχει αυτό το πολύ αυστηρό σύστημα ελέγχου και δειγματοληπτικού ελέγχου και χρειάζεται να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτό το σύστημα ελέγχου. Επίσης, όσον αφορά τον κίνδυνο που περιέχει αυτός ο έλεγχος, Πρέπει να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στο χοντρικό και στο ε, λιανικό εμπόριο και ανάμεσα στα ε, προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία. Όπως ε, είπε και ο κύριος Χόισλιν, χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος ελέγχου και φυσικά αυτό το σύστημα ελέγχου πρέπει να παραμείνει η αρμοδιότητα των εμπειρογνωμόνων και να μην ε, ενσωματωθεί σε άλλες υπηρεσίες. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όσον αφορά τους ελέγχους στις ε, τρίτες χώρες υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις ε, προδιαγραφές που τηρούνται και στα διαθέσιμα μέσα για να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι σε τρίτες χώρες, καθώς και στα διαθέσιμα μέσα επιτήρησης αυτών των ελέγχων. Σπόροι επίσης και ζωοτροφές και οι δικές μας εμπειρίες. Οι δικές μας εμπειρίες με την ε, Διεθνή Τράπεζα Σπόρων είναι πάρα πολύ καλές. Πιστεύουμε πως αυτό είναι ένα όργανο το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και χρειάζεται φυσικά διαφάνεια στη λειτουργία του. Στη δική μας επιχείρηση είμαστε, έχουμε πάρα πολύ εξειδικευμένες καλλιέργειες και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ το σύστημα αυτό. Και όσον αφορά τις ε, ζωοτροφές υπάρχουν ορισμένες Υπάρχουν ορισμένοι τομείς στους οποίους ε, χρησιμοποιούμε ζωοτροφές πρωτεϊνούχες, ζωοτροφές από συμβατικές τιμές, αλλά υπάρχει ολόνα και αυξανόμενο ενδιαφέρον για βιολογικές ε, πρωτεϊνούχες ζωοτροφές. Για παράδειγμα, βιολογική σόγια. Και υπάρχει ένα όριο 5% ε, εξαίρεσης 5% σε βιολογικές ζωοτροφές, το οποίο πιστεύουμε πως πρέπει να αλλάξει. Και γι' αυτό χρειάζονται προγράμματα, ερευνητικά προγράμματα τόσο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επίσης η τελευταία ερώτηση που μας ε, τέθη ήταν αν έχουμε ανησυχίες σχετικά με τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Οι βιολογικοί κτηνοτρόφοι φυσικά χρειάζεται να γνωρίζουν τι ε, ζωοτροφές δίνουν στα ζώα τους και πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ποια είναι η διαδικασία παραγωγής αυτών των ε, ζωοτροφών και ποια η διαδικασία του ελέγχου για το εάν είναι βιολογικές ή όχι. Όλα αυτά είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι πάρα πολύ σημαντικά και αποφασιστικά στοιχεία για τον χαρακτηρισμό ε, ενός προϊόντος ε, ως βιολογικό. Και φυσικά χρειάζονται κανόνες και ρυθμίσεις οι οποίες πολλές φορές πρέπει να γίνουν ε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως χρειάζεται έλεγχο σε κάθε περίπτωση για το αν το πεδίο εφαρμογής είναι το κατάλληλο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, περιέχει έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό πράξεων κατά εξουσιοδότηση, χωρίς όμως να αποσαφηνίζει πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τον έλεγχο, σχετικά με τα όρια και το πεδίο των αρμοδιοτήτων. Κυρίε και κύριοι, η συζήτηση για αυτόν τον νέο κανονισμό μας δείχνει ότι όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο περισσότερες εξελίξεις, τόσο περισσότερη έρευνα χρειάζεται. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο έχουμε σήμερα και στο οποίο κινούμαστε για την βιολογική γεωργία, το οποίο μπορούμε να ε, βελτιώσουμε. Και εάν χτίσουμε πάνω σε αυτό το υφιστάμενο πλαίσιο, τότε μπορούμε να αποφύγουμε πάρα πολλέ ε, περιπτώσει ε, νομικής ε, ασάφειας. Διότι αυτή η ασάφεια υπάρχει ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλες τις διαφορετικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες και σαφείς προτάσεις για την μεταρρύθμιση του κανονισμού και θα, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τα θεσμικά όργανα να τις ε, λάβουν σοβαρά υπόψη, ιδιαίτερα όσον αφορά την επεξεργασία, το εμπόριο των βιολογικών προϊόντων και το μοντέλο της ε, μελλοντική βιολογικής οικονομίας. Σας ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στον δεύτερο καλεσμένο πυρογνώμονά μας. και μετά θα γίνουν ε, ερωτήσεις. Θα έχουμε και δεύτερο μέρος ε, στη δημόσια Ακρόαση, με άλλους τρεις εμπειρογνώμονες. Στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης θα προηγούνται όσοι δεν έλαβαν μέρος ε, στη συζήτηση του πρώτου τμήματος, για να μπορέσουμε όλοι να λάβουμε το λόγο. Περνάμε στο δεύτερο μας εμπειρογνώμονα, τον κύριο Γιούρν Σάντερς, που είναι ερευνητής στο Ομοσπονδιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τις Αγροτικές Ζώνες, για την δασοκομεία και την αλία στη Γερμανία. Παρακαλώ κύριε Σάντερς, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την σημερινή πρόσκληση στην ακρόαση αυτή και για τη δυνατότητα να παρουσιάσω ορισμένες παρατηρήσεις από την προοπτική και από, την οπτική γωνία ενός επιστημονικού πολιτικού συμβούλου. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και αξιολόγησης ε, με πολλούς ε, συναδέλφους μου. Κάναμε μία εξπόστα αξιολόγηση του κατά πόσο οι υφιστάμενοι κανόνες είναι αποτελεσματικοί και του πώς μπορούμε να επιτύχουμε το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα για τον κανονισμό. Πρέπει να κοιτάξουμε προς το μέλλον και το ενδιαφέρον μας, το συμφέρον μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για την βιολογική γεωργία έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσοστό βιολογικών καλλιεργειών τα επόμενα χρόνια. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα. Ταυτόχρονα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι οι ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόνο ένα από τα μέσα ενίσχυσης της ε, βιολογικής ε, γεωργίας στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα επίσης της ε, στήριξης, της έρευνας, της επικοινωνίας. Θεωρώ πως εάν θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο της αύξησης της βιολογικής γεωργία στην Ευρώπη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να, ε, να λάβουμε υπόψη και τα υπόλοιπα συνοδευτικά μέτρα, να κάνουμε μια ενδελεχή ανάλυση των ε, ε, λόγων έτσι, και των αιτιών έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια σωστή συνεκτική πολιτική σχετικά με την οικολογική και βιολογική γεωργία. Χρειάζεται μια συνεκτική πολιτική και ενιαία πολιτική σε όλον τον ευρωπαϊκό χώρο. Επίσης κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι για να αυξηθεί και να ενισχυθεί η βιολογική καλλιέργεια στην Ευρώπη χρειάζεται ενίσχυση και χρειάζεται αύξηση των ε, φορέων που εργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό. Επίσης είναι κατανοητό ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, προσπαθούν να λάβουν υπόψη και το ε, ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και το εθνικό δίκαιο που ισχύει σε κάθε χώρα. Όμως θα ήθελα να αναρωτηθούμε εάν πραγματικά πρέπει να εστιάσουμε στο δίκαιο και όχι σε μια στρατηγική δημιουργία ενός ε, πλαισίου. Ενός πλαισίου το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα από τη μία να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ε, πρωτοβουλίες, πρωτοβου... Ε, πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα μπορέσουν να μας οδηγήσουν για παράδειγμα σε μια αλλαγή του πλαισίου, μια τροποποίηση του πλαισίου και από την άλλη να έχουμε στη διάθεσή μας τις αναγκαίες πληροφορίες, τα αναγκαία στοιχεία έτσι ώστε να ε, το δρομολογήσουμε. Και γι' αυτό χρειάζεται φυσικά ε, ενίσχυση της έρευνας και της ε, ανάπτυξης. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική η επικοινωνία και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με τους φορείς που ασχολούνται με αυτή την έρευνα και την ανάπτυξη στον κλάδο της βιολογικής καλλιέργειας. Πρέπει να δούμε τι στόχους έχει η βιολογική γεωργία και σε όλη την επικράτεια της Ένωσης και στα εθνικά κράτη και στις περιφέρειες μεμονωμένα. Επίσης, πρέπει να δούμε τι θέλουμε να πούμε με την ανάπτυξη, τι θέλουμε να πούμε με την εξέλιξη και τι θέλουμε να πούμε με την επέκταση της φιλολογικής γεωργίας. Τον Μάρτιο δημοσιεύτηκε η πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που ήταν αντικείμενο πάρα πολύ δημιας κριτικής. Στη Γερμανία η κριτική εστίασε, πρώτα στις πράξεις κατά εξουσιοδότηση, που ήταν το μαύρο κουτί της ε, του όλου κανονισμού, από την άλλη οι εξαιρέσεις και, για, και ε, το τρίτο σημείο ήταν οι οριακές τιμές για το χαρακτηρισμό ενός προϊόντος ως βιολογικό. Η βιολογική γεωργία έχει ως θεμελιώδη αρχή ε, την ε, όσο το δυνατόν αποφυγή των συμβατικών εξωτερικών συστατικών. Και εάν εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, τότε αυτά τα εξωτερικά συστατικά πρέπει να είναι ε, και εκείνα βιολογικά. Τώρα, το θέμα είναι, θέλουμε να δεσμευτούμε και να προσπαθήσουμε για να ακολουθήσουμε αυτε, αυτόν τον κανόνα ή όχι. Και πρέπει να κατανοήσουμε και να αποδεχτούμε το ότι οι φυστάμενοι κανόνες είναι αρκετά αδύναμοι για να γίνει αυτό. Υπάρχουν αυτές οι, αυτές οι εξαιρέσεις οι οποίες δυστυχώς έχουν γίνει κανόνα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, σπόροι. Στην Μεγάλη Βρετανία ανάμεσα στο 2007 και το 2011 είχαμε αύξηση αυτών των εγκρίσεων κατά εξαίρεση κατά πολύ μεγάλο ποσοστό για, τα, ε, για το σιτάρι ενώ υπήρξε μείωση τη συνολική καλλιέργεια σιτηρών κατά 11%. Αυτές οι εξελίξεις είναι κατά ένα σημείο κατανοητές, διότι τα συμβατικά προϊόντα κοστίζουν λιγότερο και οι φορείς που τα ε, διαθέτουν στην αγορά δεν έχουν αρκετά κίνητρα για να αλλάξουν την καλλιέργεια αυτή σε βιολογική. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από ε, διαφορετικότητα. Για παράδειγμα, διαφορετικότητα στην διαθεσιμότητα των σπόρων. Και αυτή η πολυμορφία στην Ευρώπη είναι, είναι επίσης σημαντικό να δούμε ότι οφείλεται και στις ε, εδαφικές ε, και στις γεωγραφικές διαφορές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση στις περιφέρειες και στους ε, περιφερειακούς φορείς και στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας. Διότι εάν θέλουμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο χρειάζεται μεγαλύτερη πίεση προς αυτούς τους φορείς. Μεγαλύτερη πίεση ώστε αυτοί οι φορείς να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και πρέπει επίσης να προσέξουμε αυτή η πίεση να μην οδηγήσει σε δυσανάλογα αρνητικά αποτελέσματα. Δηλαδή, χρειάζεται μία προσπάθεια εξισορρόπησης, να δούμε πώς να, έχουμε αρκετή πίεση αλλά όχι υπερβολική. Τώρα, όσον αφορά τις ε, εξαιρέσεις στην έγκριση, εδώ πρέπει να δούμε επίσης τις ε, διαφορές ε, των, διάφορων, των διάφορων τύπων επιχειρήσεων και πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να διασφαλιστεί το 100% της βιολογικής προέλευσης. και να δοθεί επίσης έμφαση στα τοπικά βιολογικά προϊόντα, στα πρωτε, σε πρωτεϊνούχες ε, ζωοτροφές και για γιατί συγκεκριμένα, αν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το 100% βιολογική προέλευση, πρέπει να περιμένουμε ότι η αγορά δεν θα αντιδράσει τόσο γρήγορα όσο το επιθυμούμε και πως υπάρχουν άλλες αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η αγορά της Ασίας για παράδειγμα, η οποία έχει την δυνατότητα να αντιδράσει ταχύτερα από εμάς. Επίσης, αυτό το 100% σημαίνει επίσης και επιπρόσθετο κόστος και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντέξουμε αυτό το κόστος και πώς θα μπορέσουμε να πληρώσουμε αυτό το επιπρόσθετο κόστος. Χρειάζονται λοιπόν ειδικοί οι οποίοι θα μπορέσουν να απαντήσουν σε αυτές τις λεπτομερείς ε, ερωτήσεις. Τώρα, αν θέλουμε να καταργήσουμε αυτές τις ε, εξαιρέσει τις άδειες ε, για εξαίρεση. Αυτό θα έχει και αρνητικές επιπτώσεις και οι αρνητικές επιπτώσεις ε, ε, σημαίνει αύξηση της τιμής. Ωστόσο δεν είναι ακόμα σαφές το πλαίσιο, είναι πάρα πολλά σημεία τα οποία μας, μας είναι άγνωστα. Για παράδειγμα το κόστος των βιολογικών σπόρων στα διάφορα κράτη-μέλη ή το θέμα της διαθεσιμότητας βιολογικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών. Πρέπει να γνωρίζουμε το κόστος, να γνωρίζουμε τις τιμές του κάθε προϊόντος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή ανάλυση του συνολικού κόστους αυτής της ε, κατάργησης των εξαιρέσεων. Επίσης πρέπει να ε, αναλύσουμε το θέμα των επιτρεπόμενων ουσιών στα βιολογικά προϊόντα ακούγεται ότι αυτό είναι μία αλλαγή από τον έλεγχο της διαδικασίας στον έλεγχο του τελικού προϊόντος. Μία αλλαγή δηλαδή προς ανατολισμού στον έλεγχο της βιολογικής ε, γεωργίας. Εγώ έτσι όπως το καταλαβαίνω βλέπω ότι χρειάζεται καταρχάς εναρμόνιση και δεύτερον ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα. Είναι επίσης δύσκολο θέμα το θέμα της ε, ρύθμισης του ελέγχου των βιολογικών προϊόντων ακριβώς διότι υπάρχει αυτή η πολυμορφία και αυτό σημαίνει ότι 24 κράτη-μέλη έχουν 24 ε, διαφορετικούς τρόπους ελέγχου αυτών των ε, οριακών τιμών καταλήπων. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται για να διαπιστωθούν αποκλήσεις και για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάποια μόλυνση του προϊόντος από άλλα συστατικά στοιχεία πλήν των βιολογικών ή από επικίνδυνα, από κίνδυνες ουσίες. Εδώ πρέπει να αναλογιστούμε εάν αυτή η εμπιστοσύνη των καταναλωτών θα κλονιστεί μακροπρόθεσμα. Διότι αυτοί οι έλεγχοι φυσικά δεν αφορούν μόνο τα βιολογικά προϊόντα, αλλά και γενικότερα τα υπόλοιπα προϊόντα και αυτό συνδέεται άμεσα και με το ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2006 έως το 2011 για παράδειγμα, υπήρξε μεγάλη αύξηση, κατά 50% αύξηση στη ζήτηση βιολογικών προϊόντων. Προσπάθησα λοιπόν, κλείνοντας, να επικεντρωθώ σε αυτές τις δύο πτυχές και σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και με χαρά μου θα ακούσω ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Σάντερς. Έχουμε στην αίθουσα και εμπειρογνώμονες από την Κόπα Κοζέκα, τον κύριο Ρουσό και τον κύριο Γιάν Πλάγκα από την Διεθνή Ομοσπονδία Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας, την ΙΦΑΜ. Θα τους δώσω το λόγο για σύντομες παρουσιάσεις. Παρακαλώ πρώτα στον εμπειρογνώμονα από την Κόπα Κοζέκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα, μας δίνετε δυνατότητα να μιλήσουμε σε αυτό το βήμα. Εκπροσωπώ σαν παραγωγός τους παραγωγούς, τους Ευρωπαίους των βιολογικών προϊόντων και τους συνεταιρισμού και συμμερίζομαι με διαπίστωση μαζί σας, δηλαδή ότι έχουμε σημαντική αύξηση της κατανάλωσης των βιολογικών προϊόντων, ε, μία από τέλμα της μετατροπής προς βιολογικές καλλιέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αύξηση των εισαγωγών. Ε, το ερώτημα που τίθεται και στο οποίο θα θέλαμε να απαντήσουμε πρακτικά και τεχνικά είναι το εξής. Θέλουμε πραγματικά να ηγηθούμε στη βιολογική ε, για την ευρωπαϊκή κοινωνία και για την εικόνα μας στον κόσμο, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία, ενθαρρύνοντας φυσική και ποιοτική γεωργία η οποία ενισχύει και την αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών στην ποικιλομορφία τους, διότι αντιλαμβανόμεθα ότι η βιολογική ε, καλλιέργεια δεν αναπτύσσεται εξίσου σε όλες τις περιοχές. Λοιπόν, μια νέα νομοθεσία πρέπει να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Αν ναι, αν έχουμε αυτή τη φιλοδοξία και δείξαμε ότι μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα για απασχόληση, για προστιθέμενη αξία, θα πρέπει να μπορέσουμε να απευθυνθούμε προς όλους τους παραγωγούς, τους ευρωπαίους παραγωγούς ε, στις διάφορες περιφέρειες που επικύλουν. Εκπροσωπούμε περίπου 200, 205.000 ε, καλλιέργειες, αλλά μόνο 5% της καλλιεργούμενης έκτασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να επιτύχουμε μια αρμονική καλλιέργεια και επιμένω επί συγκεκριμένου σημείου πρέπει να αποφύγουμε την αύξηση των διαφορών κυρίως ε, στις πιο εντατικές ε, περιοχές που καλλιεργούνται, ε, διότι βλέπετε ότι πολλές βασικές πρώτες ύλες, κυρίως δημητριακά, σιτηρά, χρειάζονται, διότι αυξάνεται η ζήτηση στην αγορά, όσον αφορά τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα και χρειαζόμαστε όλους τους γεωργούς και να παραμείνουν οι ανοιχτέ οι πόρτες που εκείνους που θέλουν να διαλέξουν αυτή την προσέγγιση. Κυρίως σε εντατικοποίηση της γεωργίας που περιπλέκει ε, το πέρασμα προς την βιολογική γεωργία. Στο επίπεδο της κόπα κοζεκά ζητάμε να, ε, να εφαρμοστούν τεχνικές προσαρμογές υπό τη μορφή παρεκκλήσεων αλλά δεν θα πρέπει να αυτός σκοπός να είναι προσαρμογές οι οποίες συνοδεύουν την ε, ανάπτυξη επιμείναμε ευτυχής των μεικτών εκμεταλλεύσεων διότι προς εκείνη την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Επίσης θα πρέπει ε, για τα αναπαραγωγικά ζώα και για, τις, και για τους σπόρους θα πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το γενικό απόθεμα το αναπαραγωγικό. Λοιπόν, αλλάζει η κατάσταση, δεν έχουμε αποκλειστικά τέτοιο αναπαραγωγικό υλικό βιολογικό, σταδιακά αλλάζει η κατάσταση, βλέπουμε να δημιουργούνται και νέοι πόροι, νέες πηγές Θέλω να επιμείνω επί των ελέγχων. Είμαστε υπέρ των όσων προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μακρηγόρησα και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριο Πλαγκέ από την ΙΦΟΑΜ, την Διεθνή Ομοσπονδία Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για την ε, δυνατότητα που μου δίνετε να κάνω μια παρέμβαση ως εκπρόσωπος ε, της ε, βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη και της σχετικής ομοσπονδίας. Εμείς εκπροσωπούμε την βιολογική γεωργία στην Ευρώπη. Και από την αρχή ενταχθήκαμε στις διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση του κανονισμού και υποβάλαμε κάποια θέματα που θα πρέπει να τεθούν κατά προτεραιότητα ε, όπως το θέμα της εκτροφής ε, πουλερικών και ζητήσαμε μια σταδιακή διαδικασία στις ε, επαφές που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια σταδιακή διαδικασία με συμμετοχή των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των διανομέων, αλλά και των πελατών, των καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ε, κάνει μια επανάσταση στον κομμάτι των βιολογικών καλλιεργειών παρά τις ε, αντιρρήσεις όλων και χωρίς να συμβουλευτεί τους εμπειρογνώμονες. Και εμείς αυτό το αρνούμαστε. Αρνούμαστε ως ε, βιολογικοί καλλιεργητές όλη αυτή τη ριζική αλλαγή που έχει προταθεί και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μία πρόταση κανονισμού η οποία θα έχει λάβει υπόψη της και θα δώσει μία ευκαιρία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να βελτιώσει τον κανονισμό. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές απόψεις για το ε, χρονοδιάγραμμα και γιατί ε, με το φυστάμενο χρονοδιάγραμμα δεν μπορεί να επιτύχει τους ε, προσδοκόμενους στόχους αυτός ο κανονισμός και το Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει εάν αυτός ο κανονισμός μπορεί να λειτουργήσει και μπορεί να επιτύχει το στόχο του με, αυτές, με τις χιλιάδες τροπολογίες που αναμένεται να ε, υποβληθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς κάνουμε μία έκκληση ως ε, βιολογικοί αγρότες για μία σωστή και συνετή τροποποίηση του κανονισμού. Σας ευχαριστώ. Έχουμε τώρα συζήτηση. Θα υποβληθούν ερωτήσεις στους εμπειρογνωμονές μας γιατί έχουμε δημόσια κρόση και άρα θα πρέπει να μπορούμε να υποβάλουμε ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις τους 18 συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Έχουμε μόνο 1,5 λεπτό για τον καθέναν. Παρακαλώ ε, μην ε, στεναχωριέστε που σας δίνω τόσο λίγο χρόνο, αλλά δυστυχώς έχουμε πολλούς ομιλητές, πολλές ερωτήσεις και πρέπει να κάνουμε μια ορθολογική διαχείριση του χρόνου Ο κύριος Λίντς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω. Μία για τον κάθε εισηγητή. Η πρώτη ερώτηση προς τον κύριο Πίντς Τσουλιόφενστάιν έχει να κάνει με τις ε, μικτές ε, εκμεταλλεύσεις. Υπάρχουν διαφορετικές ε, διαδικασίες και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να αποφασίσει κάποιος ε, καλλιεργητής να αλλάξει τον ε, τρόπο που εργάζεται. Εσείς ε, θεωρείτε πως υπάρχουν τέτοιες εκμεταλλεύσεις οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν μεικτά με επιτυχημένο τρόπο, μπορεί να υπάρξει δηλαδή αυτή η συνύπαρξη Επίσης αναφέρθηκε το 2020-2021 ως ημερομηνία τη οποία θα επιφερεύτε στις αλλαγές εσείς. Μπορείτε να μας πείτε τις δικές σας εκτιμήσεις για το χρονοδιάγραμμα και μπορείτε να μας πείτε αν εκτιμάτε ότι μπορούν όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να το τηρήσουν. Επίσης, η δεύτερη μου ερώτηση προς τον ε, κύριο Σάντερς. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα βιολογικά προϊόντα, βιολογικά τρόφιμα στα καταστήματα και πως υπάρχει και αύξηση της συζήτησης, πως υπάρχει δηλαδή το αγοραστικό δυναμικό. Όσο να αφορά τους ελέγχους τώρα, που έχουν προταθεί Πώς μπορείτε να τους ε, αξιολογήσετε. Και επίσης κάτι άλλο ε, προς τον κύριο Λεόβενστάιν. Εσείς τι θα μας προτείνατε για, το, για την πρόταση κανονισμού ε, που έχει υποβάλει η Επιτροπή να τον αλλάξουμε, να τον τροποποιήσουμε, να τον επεξεργαστούμε τέλο πάντων ή να τον απορρίψουμε και να υποβληθεί κάποιος άλλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο Θα είμαι λακωνικός. Εγώ διαπιστώνω ότι η βιολογική γεωργία έχει αποκτήσει ένα δυναμισμό και μια δυναμική που καλό θα ήταν να μην την αναχαιτήσουμε. Και θα πρέπει ο κανονισμός αυτό το στόχο να ε, υλοποιήσει και να υιοθετήσει μια διασταλτική ερμηνεία της βιολογικής γεωργίας, γιατί είναι συμβολική η εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας των γενικών εξελίξεων που διαπιστώνουμε στην κοινωνία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να προβληματιστούμε ε, για να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε για ολόκληρη τη γεωργία μας. Το είπατε. Θα πρέπει λοιπόν να διαρωτηθούμε τι ε, μοντέλο ανάπτυξης θέλουμε για τη γεωργία μας. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε τις σωστές ερωτήσεις στη συζήτηση. Είπατε ότι η βιολογική γεωργία έχει τεράστιο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία νέων θεμελίων ε, στη γεωργία προκειμένου να γίνει ανταγωνιστική και αηφόρος. Μιλήσετε για την προσφορά στη δημόσια υγεία, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ε, στην ε, δημιουργία μιας νέας στρατηγικής. Και δεν θα πρέπει να φέρουμε αντιμέτωπη στη συμβατική γεωργία με τη βιολογική, αλλά να τις θέσουμε ως συμπληρωματικέ. Και επίσης να έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα ε, ο χρονικός ορίζοντας έχει βραχυπρόθεσμο, μέσο και μακροπρόθεσμο στάδιο. Θα πρέπει όλες αυτές τις πτυχές να τις λάβουμε υπόψη. Αυτό που λείπει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο ορισμός της βιολογικής γεωργίας. Γιατί ε, αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αν θέλουμε κοινό στόχο θα πρέπει να έχουμε μια κοινή αφετηρία. Και δεν φαίνεται ο στόχος μεταξύ ε, του εδάφους, ε, της χλωρίδας και της πανίδας, ε, των φυτών και των ζώων. Αυτά είναι απαραίτητες προϋποθέσεις δεδομένων των ανησυχιών που έχουν τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έκαναν τις παρουσιάσεις. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις που έγιναν. Πιστεύω ότι το σημαντικότερο όλων είναι ότι η μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει να ενθαρρύνει τον κόσμο να κινηθεί ε, τώρα περισσότερο από ό,τι κατά προς τη βιολογική γεωργία. Δεν υπάρχουν αρκετά βιολογικά προϊόντα που προσφέρονται. Για τον κύριο Βεν Λεβενστάιν θα ήθελα να ρωτήσω πώς από πλευράς ε, των παραγωγών βλέπουν την αξιολόγηση του κινδύνου. Πώς θα βοηθήσει η αξιολόγηση του κινδύνου. Δεν θα σημαίνει ότι θα αυξηθεί πολύ η γραφειοκρατία. Δεν σημαίνει ότι κινούμαστε πολύ μακριά. Κάνουμε υπερβολικά πράγματα. Ίσως ε, δεν θα δεν υπάρχουν αρκετοί που θέλουν να αγοράσουν, δεν θα θέλουν πολλοί μεσάζοντες να αγοράζουν βιολογικά προϊόντα αν συμβεί αυτό. Και ίσως δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα για τις μικρές και πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις και τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τι θα συμβεί. Τι συμβαίνει πριν τελικά να φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων τα βιολογικά προϊόντα. Τι παρεμβάλλεται. Αυτές οι πτυχές λοιπόν πώς θα αντιμετωπιστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα οι μεικτές εκμεταλλεύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εκμεταλλεύσεις ίσως είναι μεγαλύτερες από ό,τι αλλού και πολλές, πολλοί γεωργοί παράγουν βιολογικά προϊόντα, μείωσαν την παραγωγή, δεν μπορούσαν να πουλήσουν τα προϊόντα τα τελευταία χρόνια και τώρα έχουν ένα δίλημα. Δηλαδή διπλασιάζουμε ή τα παρατάμε ή θα βάλουν και την άλλη μισή εκμετάλλευση να παράγει βιολογικά προϊόντα, είναι πολιτική απόφαση, θα έχουν κάποια επιδόματα για την αλλαγή. Ή τελικά θα κατηγορηθούν κάποιοι που παίρνουν τα επιδοτήματα χωρίς, τις τα επιδοτήματα χωρίς τελικά να κάνουν την αλλαγή θα πρέπει να επιτρέψουμε τις μεικτές εκμεταλλεύσεις. Τώρα όσον αφορά τους σπόρους έχουμε περασμένους ε, πόρους. Δεν θα πρέπει τελικά κάποιος γεωργός να μην μπορεί να παράγει κάτι βιολογικά προϊόντα, λείπουν οι σπόροι. Θα... Είναι σκάνδαλο αυτό. Κανόνα θα πρέπει να είναι. Ε, όταν μπορεί να λέξει την κατάσταση ο γεωργός που παράγει βιολογικά προϊόντα θα πρέπει τελικά να λάβει το σπόρο και να κάνει τη βιολογική καλλιέργεια. Για τις ζωοτροφές οι ζωοτροφέ θα πρέπει να παράγονται από τον καλλιεργητή που παράγει βιολογικά προϊόντα για να τρέφει τα ζώα του. Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, θα πρέπει να αγοράσει μη οργανικά τρόφιμα και να πωλήσει τα ζώα ως έχουν. Τουλάχιστον παράγεται ένα είδος ε, τρόφιμο με αυτόν τον τρόπο. Και τέλος θέλετε να αλλάξετε τον, καιρό, αν το αμφισβητώ. Κοιτάξτε τι γίνεται. Λοιπόν, οι μη οργανικοί καλλιεργητές πώς ελέγχουν ε, παράγουν πολύ λίγο διοξίδιο το, το άνθρακος. Και τελικά η άλλη παραγωγή, παραγωγή ε, γίνεται τελικά με μηχανικά προϊόντα και τελικά παράγουν πάρα ε, πολλά αέρια του θερμοκηπίου άμα χρησιμοποιούνται περίπλοκοι τρόποι καλλιέργειας των προϊόντων και παράγουμε αέρια. Ευχαριστώ. Κύριος Κούσμιουκ. Και οι δύο εμπειρογνώμονες δεν επέκριναν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενώ άλλοι συνάδελφοι είπατε ότι είναι τόσο φιλόδοξες οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το παρατραβάν τόσο πολύ που όχι μόνο δεν θα προαγάγουν την βιολογική γεωργία αλλά θα την περιορίσουν. Αυτή είναι η άποψη των Ευρωβουλευτών ενώ οι εμπειρογνώμονες δεν αντιτάχθηκαν στην πρόταση. Το θέμα είναι ότι έχουμε γύρω στις 225.000 ε, ε, βιολογικές εκμεταλλεύσεις, ε, ένα μικρό τμήμα της συνολικής γεωργικής παραγωγής. Οπότε οι υπάρχουσες νομοθετικές διατάξεις φαίνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα πρόσφορες και ευνοϊκές για τη βιολογική γεωργία, εξού και το χαμηλό της μερίδιο σε σχέση με το σύνολο της γεωργίας. Ο κύριος Λεβενστάιν μίλησε για την ανάγκη κατάργησης των μεικτών καλλιεργειών. Και μάλιστα ανέφερε το 2021 ως ε, προθεσμία. Σε μερικές περιοχές όμως διαπιστώσαμε ότι το 40% περίπου των βιολογικών καλλιεργειών είναι μικτές καλλιέργειες. Οπότε αν θέσουμε τέτοιους όρους ε, και την δυνατότητα κατάργησης θα επηρεάσει αρνητικά την βιολογική παραγωγή θα την περιορίσει, κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έρτοκ. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνεται να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τους ε, βιολογικούς καλλιεργητές ε, θα πρέπει εκείνοι να έχουν κάποια ωφέλη να είναι θετικές οι συνθήκες και να μην αυξάνεται το βάρος επάνω τους. Έτσι θα πρέπει να κινηθούν οι κανονισμοί, διότι οι βιολογικές καλλιέργειες αυξάνονται με δυναμικό τρόπο ε, και θα πρέπει να τεθεί το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο κύριος Λεβενστάιν ανέφερε ότι το παρόν πλαίσιο λειτουργεί σωστά. Θα μπορούσε κανείς λοιπόν να διαρωτηθεί αν έχει νόημα να θεσπίσουμε ένα νέο κανονισμό ή αν είχε νόημα ε, να παρατήσουμε την παράλληλη καλλιέργεια μετά από πλευράς ασφαλείας των τροφίμων. Θα έπρεπε να απαγορευτούν οι απλοί σπόροι εντελώς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις έχω όσον αφορά το πρόβλημα των οριακών τιμών λέει ο κύριος Γιάρ. Μήπως έχουμε χάσει την ευκαιρία να ορίσουμε αυτέ, τα όρια αυτών των ε, τιμών. Επίσης, ο προσανατολισμός μας αλλάζει ανάλογα με το αν ένα προϊόν είναι βιολογικό ή όχι. Επίσης, ε, το, όσον αφορά τα, τις βλαβερές ουσίες που βρίσκονται ε, στα προϊόντα, ίσως θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τις επιδοτήσεις για τον έλεγχο αυτών ε, των ε, προϊόντων. Τώρα, εσείς κύριε Λόβενσταν είπατε ότι υπάρχει ένας προσανατολισμός ε, ως, προ, και μια εστίαση στην διαδικασία. και μιλήσατε επίσης για αυτές τις εμικτές εκμεταλλεύσεις, για το, τα πρωτεϊνούχα, τις πρωτεϊνούχες ζωοτροφές και θα ήθελα λοιπόν εγώ να σας ερωτήσω εσείς. Έχετε σκεφτεί τι θα μπορούσε να γίνει με τη μεταβατική περίοδο και το χρονοδιάγραμμα ε, για, αυτές, ε, αυτή τη μετάβαση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Έριξον. Σας ευχαριστώ. Στην πατρίδα μου έχουμε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που επικρατεί και σε άλλες χώρες. Έχουμε μια αύξηση, εντυπωσιακή αύξηση της ζήτησης των βιολογικών προϊόντων και άρα και μια άνθηση της βιολογικής γεωργίας. Όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται για τον κλάδο αυτό. Οπότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι αναγκαία αυτή η τροποποίηση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά πόσο θα είναι υποφελής. Θα πρέπει πρώτα να κάνουμε μια σωστή επισκόπηση της κατάστασης και να λάβουμε υπόψη ότι δεν έχουν ακόμη κερδίσει τα βιολογικά προϊόντα την εμπιστοσύνη των ε, καταναλωτών. Αυτό είναι το επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος όλο και περισσότερο ενδιαφέρεται και ζητά ε, βιολογικά προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα σύστημα ελέγχου που θα ικανοποιεί και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές και φυσικά ε, θα είναι και αποτελεσματικός. Μία μικρή ποσότητα φυτοφαρμάκων της γειτονικής παραγωγής μπορεί να καταστρέψει την ε, βιολογική καλλιέργεια με ανεπανόρθωτες συνέπειες για το εισόδημα του βιοκαλλιεργητή. Θα πρέπει να επιδιώξουμε το σύστημά μας να είναι αποτελεσματικό και όχι προβληματικό που θα κλονίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και θα οδηγήσει σε χρεοκοπία τους ε, βιοκαλλιεργητές. Ναι. Ρίξτε μια ματιά και στη Βόρεια Ευρώπη δεν έχουμε αρκετούς ε, βιοκαλλιεργητές για να καλύψουν την ανάγκη τη ζήτηση σε βιολογικά προϊόντα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να περιορίσουμε ακόμη περισσότερο τη βιολογική γεωργία. Η κυρία Ράνς Γκαρσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονές μας. Η Ισπανία έχει ηγετική θέση στην ε, βιολογική παραγωγή της Βιολογικής Ένωσης. Γι' αυτό θέλουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω την κατάσταση, να ενισχύσουμε την κατανάλωση. Το 40% των ε, ισπανικών ε, καλλιεργιών είναι μικτές και ουδέποτε δεν εντοπίστηκε ε, περίπτωση απάτης. Μπορεί πολιτικά, οικονομική να είναι η ενιαία παραγωγή, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα οδηγήσει σε εξολόθρευση ένα μεγάλο τμήμα των ισπανικών καλλιεργιών. Επίσης, ε, η αγορά ζωοτροφών που δεν είναι βιολογικές ή δεν προέρχονται από την περιοχή που γίνονται οι αγορές. Σε θερμές ζώρες όπως είναι ε, της Ισπανίας, σε μια τέτοια υποχρέωση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα Μήπως ε, είναι καλύτερο να βελτιώσουμε και να διευκολύνουμε τους, ε, τους παραγωγούς χωρίς όμως ε, περιορισμούς και παράλογες απαγορεύσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Μόη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά τον τομέα των βιολογικών προϊόντων οι έλεγχοι δεν είναι αποτελεσματικοί και μέχρι τώρα πολλοί γεωργοί, πολλές εταιρείες το εκμεταλλεύτηκαν αυτό και οι δηλώσεις που έκαναν για να πετύχουν τη χρηματοδότηση πολύ συχνά ήταν ψευδείς και αυτό έχει αποκρυφτεί από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ζητώ λοιπόν να βελτιωθεί το σύστημα των ελέγχων ούτως ώστε μετά να δίδονται ε, τα χρήματα για τις διάφορες επιδοτήσεις από, τα, από τον προϋπολογισμό της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και για τη λακωνικότητά σας. Ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις που έκαναν και για την εμπειρία που μας μεταδίδωσαν η βιολογική παραγωγή σήμερα ε, αποτελεί με τις προσδοκίες του καταναλωτού. Και αυτό που θα πρέπει να θεωρήσουμε σαν πρόκληση είναι πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Θα πρέπει οι κανόνες να εφαρμόζονται στις διάφορες χώρες με έναν τρόπο παρόμοιο και ο καταναλωτής από όπου και να προέρχεται το προϊόν να έχει τη βεβαίωση ότι αυτό που αγοράζει είναι αυτό που αναφέρεται στην ετικέτα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να έχει ο δημόσιος τομέας τη δυνατότητα του ελέγχου, θα πρέπει αυτή η δυνατότητα ελέγχου να, να εφαρμόζεται από τους διάφορους οργανισμούς πιστοποίησης, ε, αλλά θα πρέπει να είναι αυστηρός ο έλεγχος. Η αυστηρότης ε, επιτρέπει εν συνεχεία ε, να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη και αυτή η εμπιστοσύνη αφορά εδρεύει επί των εκμεταλλεύσεων, των εκμεταλλεύσεων που έχουν και βιολογικές καλλιέργειες και παραδοσιακές καλλιέργειες και θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε μικτές εκμεταλλεύσεις αν θέλουμε να έχουμε πραγματική ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας στην Ευρώπη. Διότι ανάλογα με τη γεωγραφική θέση, καμιά φορά είναι δυνατόν σε μια εκμετάλλευση να υπάρχει μία, να υπάρχει μία ή δύο βιολογικές καλλιέργειες, αλλά να μην είναι πλήρης όλη η παραγωγή βιολογική. Τέλος, θα πρέπει να τηρηθεί η δυνατότητα παραγωγής, βιολογικής παραγωγής, να προστατευθεί η βιολογική καλλιέργεια δυνατότητα, να μην κλειστεί από παντού, να περιοριστεί ε, και τελικά να είναι ασφικτικός ο κλειός που θα δημιουργηθεί γύρω της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Γλέζος. Παρακαλώ. Ερωτήσεις. 1,5 λεπτό έχετε κύριε Γλέζο. Αξιόλογες εισηγήσεις όμως παρέλειψαν τον τομέα τον νησιωτικό. Και το πρώτο μου ερώτημα είναι γιατί. Πριν 40 χρόνια, όντας Ευρωβουλευτής, βοήθησε να δημιουργηθεί ειδική επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα νησιά. Καταργήθηκε αυτή η επιτροπή, όμως τα νησιά υπάρχουν. Και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ένα γεγονός, ότι όντως στα νησιά υπάρχει και λειτουργεί η βιολογική καλλιέργεια. Χρησιμοποιούν και την αμυψισφορά και την αγρανάπαυση και τα ζωικά λοιπάσματα. Όμως τα νησιά δεν είναι το ίδιο σε όλη την Ευρώπη. Από τις 28 χώρες μόνο 4 χώρες δεν έχουν νησιά. Και είναι άλλα τα νησιά τα, στην Ατλαντική περιοχή, άλλα τα νησιά της Μεσογείου και μέσα στη Μεσόγειο άλλα τα νησιά. Στην πατρίδα μου με τις εκατοντάδες στα νησιά υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα. Σκεφτείτε ότι εμείς δεν έχουμε χωράφια και κατασκευάζουμε χωράφι. Το, το χώρο που έχει το Προεδρείο σας είναι ένα χωράφι και αν το μισό από όλη αυτή την αίθουσα δεν το λέμε απλώς χωράφι, το λέμε χωράφα και κουβαλάμε χώμα με αναβαθμίδες να φτιάξουμε χωράφια πρόβλημα που δεν υπάρχει στα άλλα μέρη. Και επίσης επειδή δεν έχουμε νερό περιμένουμε από την έξατμισιο διαπνοή να έρθει ο κατσιφόρας όπως λέμε, να έρθει η πυκνή ομίχλη να εμπλουτίσει το φυτό με νερό. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε το καινούργιο αυτό πρόβλημα το νησιωτικό. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pan... ευχαριστώ. Ο Bogowicz. Χαίρετε. Πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα που συζητούμε. Προσοχή να μην ε, μειώσουμε την τάση που υπάρχει για μεγαλύτερη κατανάλωση των προϊόντων. Αυτή ισχύει και για τη Σλοβενία Έχουμε κάποιες παρατηρήσεις για την πιστοποίηση, για τις πιστοποίησεις. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα όρια που τίθενται των 5 εκτάριων. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ 5 ε, εκταρίων αν χρησιμοποιούνται για βοσκή ή αν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οποροκυπευτικών. Όσον αφορά τις ε, μικτές καλλιέργειες, προτείνουμε μία παράταση της δυνατότητας μια επιχείρηση να έχει μικτές καλλιέργειες, να έχουμε πιο ευρύ χρονοδιάγραμμα. Το 2021 δεν είναι πολύ κοντινό, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και αυστηρότερους ελέγχους για να μην μειωθεί η εμπιστοσύνη σε αυτά τα προϊόντα. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να συνεπιφέρει αύξηση του βάρους του διοικητικού και του οικονομικού για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τους ελέγχους για εκείνους που πουλούν ε, ε, προϊόντα προσυσκευασμένα και τα παράγουν εκείνοι αυτοί οι έλεγχοι σε αυτούς τους εμπόρους ε, αντιπροσωπεύουν υπερβολικό διοικητικό άχθος κατά την μου και θα επιβραδύνει τη διάδοση των βιολογικών προϊόντων. Ευχαριστώ. Κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ. Ε, Έχω κάποιε ερωτήσει. Προ του εμπειρογνώμονε, του οποίου και συγχαίρω θερμά, γιατί μα διαφωτίζουν για πολλά σημεία και λύνουν πολλέ απορίε μα. Εγώ κατάγομαι από την Ανταλουσία, μια περιφέρεια στην Νότια Ισπανία. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η τοπική κυβέρνηση Ανταλουσίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα στη βιολογική γεωργία και μάλιστα έδωσε και κρατικές επιδοτήσεις για τη στροφή προς τη βιολογική καλλιέργεια των παραδοσιακών, των συμβατικών καλλιεργιών. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό μεικτών καλλιεργιών και μάλιστα το τμήμα της βιολογικής γεωργίας ε, οφείλεται σε κρατικές ενισχύσεις. Έτσι είχαμε μια αύξηση του ενδιαφέροντος ε, των ε, γεωργών. Οπότε αν μας περιορίσετε τις μικτές καλλιέργειες ή τις απαγορεύσετε, σίγουρα θα εμποδίσετε την ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας στην Ανδαλουσία. Α μην ξεχνούμε ότι η κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τετραπλασιάστηκε, ενώ η παραγωγή απλώς διπλασιάστηκε. Θα πρέπει να αυξήσουμε λοιπόν την παραγωγή για να καλύψουμε τη ζήτηση. Συγκεκριμένη ερώτηση τώρα. Τι γνώμη έχετε για το γεγονός ότι για την απέτηση να υποβάλλονται όλοι οι καλλιεργητές σε σύστημα περιβαλλοντικού ελέγχου. Όχι μόνο η πρωτογενής παραγωγή, αλλά ολόκληρη η αλυσίδα να υποβάλλεται σε περιβαλλοντικούς ελέγχους. Ποια είναι η γνώμη σας για την πρόταση αυτή. Επίσης, ό,τι αφορά την ανάγκη εναρμόνισης ε, όλων των νομοθετικών διατάξεων. Ο κύριος Σάντερς αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιφερειών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κέστιγκερ θα λάβει τώρα το λόγο και κατόπιν θα ξαναδώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας για να απαντήσουν και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, κύριε Λόβενστάιν, μου έκανα μεγάλη έκπληξη αυτό που είπατε για τα διαφορετικά κριτήρια που επικρατούν Εμείς ε, οι, οι βιολογικοί καλλιεργητές έχουν πάρα πολύ υψηλά ε, πρότυπα παραγωγής και είναι πιστεύω λάθος ο τρόπος που ακολουθείτε. Εμείς πρέπει να ε, στηρίξουμε τους βιολογικούς καλλιεργητές στην Ευρώπη, διότι οι, δικοί μας, οι δικές μας προδιαγραφές είναι πάρα πολύ πιο αστηρές από τις τρίτες χώρες. Επίσης μου έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη ότι τα βιολογικά τρόφιμα πρέπει, όπως ακούγεται, να γίνουν φθηνότερα. Πιστεύω πως εδώ υπάρχει ο κίνδυνος του ντάμπινγκ των τιμών και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Επίσης μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τόσα τρόφιμα στην Ευρώπη που πετιούνται επειδή δεν καταναλώνονται. Και μην ξεχνάμε ότι το, τα φτηνά τρόφιμα σημαίνει και σπατάλη τροφίμων, σημαίνει και ότι θα υπάρχουν τρόφιμα τα οποία θα, πετάξουμε, θα καταλήξουν στα σκουπίδια. Επίσης, δεν αναφέρθηκε τίποτα για την ε, διαθεσιμότητα των ε, τροφίμων των βιολογικών τροφίμων στον ε, κανονισμό. Επίσης θα ήθελα να πω ότι η αγορά των βιολογικών σπόρων είναι πολύ συγκεντρωμένη σε συγκεκριμένες μεγάλες πολυεθνικές. Γι' αυτό λοιπόν τι συμβαίνει με αυτήν την ε, περίπτωση. Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος ε, βιολογικός πόρος πρέπει να αναγκαστεί κάποιος ε, κατατηλεργητής να καταφύγει στους συμβατικούς. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις δυσάρεστες περιπτώσεις. Μάλιστα. Τρία λεπτά έχει ο κάθε εμπειρογνώμονα μας για να απαντήσει στις ερωτήσεις και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Τρία λεπτά δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση. Δύο. Πέντε. Καλά. Ευτυχώ, ευτυχώ, Πέντε λεπτά. Λοιπόν, αξιολόγηση κινδύνου. Λογικό είναι στη διαδικασία ελέγχου να βλέπουμε εάν υπάρχει ε, κάποιος ε, μεγάλος κίνδυνος. Ε, για παράδειγμα, αν υπάρχει ένα μια μεγάλη εκμετάλλευση, κτηνοτροφική εκμετάλλευση πουλερικών εκεί πέρα είναι διαφορετικός ο κίνδυνος από τις, ε, μια πιο μικρή εκμετάλλευση. Δεν έχει νόημα ένας μικρός καλλιεργητής που καλλιεργεί βιολογικά προϊόντα να έχει τον ίδιο αυστηρό έλεγχο με έναν ε, μεγαλοκτηνοτρόφο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μεγάλη διαφοροποίηση και φυσικά πρέπει να αποφύγουμε να καταλήξουμε σε γραφειοκρατικό μολόχ. Έπειτα, να πω ότι έχω απόλυτο σεβασμό στην ε, κριτική ικανότητα των καταναλωτών. Οι καταναλωτές έχουν επίγνωση του τι σημαίνει βιολογικό προϊόν. Έχουν επίγνωση του τι συνεπάγεται ένα βιολογικό προϊόν που έχουν στο τραπέζι τους και ξέρουν πάρα πολύ καλά τι αγοράζουν, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι περιέχει ένα βιολογικό προϊόν και ένα συμβατικό προϊόν. Μην θεωρείτε τους καταναλωτές χαζούς. Τώρα, ε, μικτές εκμεταλλεύσεις. Κάποιος είπε, αν δεν κάνω λάθος, ότι μέχρι το 2020-2021 πρέπει να έχει τελειώσει αυτό το θέμα, να έχουν καταργηθεί. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Εγώ προσπάθησα να σας παρουσιάσω το, τι, ε, το πώς έχει η κατάσταση στη Γερμανία. Εμείς προσπαθούμε να καταργήσουμε αυτές τις μικτές εκμεταλλεύσεις. Τώρα, αν θα καταφέρουμε να το πετύχουμε και αν θα καταφέρουμε να έχουμε και κάποιες εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, είναι κάτι άλλο. Επίσης, ε, ένα σχέδιο ε, χρειάζεται, ένα πολυετές σχέδιο για αυτήν την σταδιακή μετάβαση. Εμείς ε, βέβαια έχουμε τις δικές μας ε, απαιτήσει στη Γερμανία για το πώς πρέπει να γίνονται αυτές οι, να γίνονται αυτές οι βιολογικές ε, εκμεταλλεύσεις. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να είναι έτσι και για τους υπόλοιπους. Απλά αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να, ληφθεί υπόψη, να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι. Γι' αυτό και γι' αυτό ε, πρέπει να οδηγηθούμε σε μια σωστή βιολογική καλλιέργεια. Δεν μίλησα όμως για καμία καταληκτική ημερομηνία κατάργηση των μεικτών εκμεταλλεύσεων. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι να κάνω μία έκκληση για να δοθούν κίνητρα για να καταργηθούν αυτές οι μεικτέ εκμεταλλεύσεις. Τώρα, ερωτήθηκα επίσης ε, μάλλον υπόθηκε ότι άσκησα μια κριτική στην πρόταση. Όχι, όχι, όχι. Και δεν το λέω αυτό το όχι επειδή θέλω να είμαι διπλωμάτικος. Απλά, ο κανονισμός έχει πάρα πολλά ε, κομμάτια και οι βιολογικές και τα βιολογικά προϊόντα αντιμετωπίζονται λες και ανήκουν σε κάποια... Ε, σε κάποιο μικρό θύλακα. Αυτό που είπα είναι ότι επιθυμώ να μεγαλώσει ο βιολογικός κλάδος, να αυξηθούν τα βιολογικά προϊόντα, διότι έτσι θα βελτιωθούν και οι συνθήκες. Επίσης, ερωτήθηκα για το αν είναι συνετό να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τον το, ε, το νέο κανονισμό, τη νέα πρόταση κανονισμού, ή αν είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε τον υφιστάμενο. Είναι όλα θέμα χρόνου. Εάν δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μα και δεν έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε, τότε ναι, μπορώ να σα συστήσω ότι σωστό είναι να ε, αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τον υφιστάμενο κανονισμό για τα, τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τα πράγματα όπως τα κάναμε μέχρι τώρα, διότι η οικολογική γεωργία εξελίσσεται, η τεχνολογία εξελίσσεται. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και το νομικό πλαίσιο να προσαρμοστεί σε αυτές τις εξελίξεις στο βάθος του χρόνου. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι θα ήταν για όλους πολύ πιο απλό εάν αποφεύγαμε όλα αυτά τα προβλήματα της εφαρμογής μιας νέας νομοθεσίας χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη. Τώρα, σπόροι. Οι σπόροι φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικοί και φυσικά το επιθυμητό και το ευκταίο είναι οι σπόροι να προέρχονται από ε, βιολογικές πηγές. Χρειάζονται έξυπνοι μηχανισμοί για να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις της αγοράς έτσι ώστε να διατεθούν στην αγορά περισσότεροι βιολογικοί σπόροι. Και εδώ φυσικά βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης και ανάγκη... Ε, αύξηση των, ε, των ελέγχων. Φυσικά δεν υπάρχουν εξαιρέσεις στην περίπτωση των βιολογικών ε, σπόρων και τη διάθεσή τους στην αγορά. Βλέπω όμως ότι οι διαδικτυακές πωλήσει βιολογικών σπόρων πάνε καλά. Ότι το σύστημα εδώ λειτουργεί ε, καλά και ότι ίσως μπορέσει να επικαλύψει το έλλειμμα που υπάρχει στους, ε, στον έλεγχο. Γεια, ευχαριστώ πολύ και εγώ, λέει ο κύριος Σάντερς. Θα ήθελα να είμαι σύντομος όσον αφορά τους καταναλωτές. Οι αναλύσεις μας ε, δείχνουν ότι οι καταναλωτές είναι κατευθύνονται είναι κατευθυνόμενοι, κατευθύνονται στο σούπερ μάρκετ και ξεχνάνε πάρα πολύ εύκολα. Έχω μια διαφορετική άποψη από τον ε, προλαλήσαντα. Δεν έχω στη διάθεσή μου βέβαια κάποια επιστημονική μελέτη για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και αν αυτό αποτελεί κίνδυνο να χαθεί εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Όπω σα είπα, οι δικέ μας αναλύσεις έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές έχουν μια συγκεκριμένη αντίληψη των ε, βιολογικών προϊόντων, όμως ε, αυτή μπορεί να διαφέρει από την πραγματικότητα. Δεν έχουν επιστημονικές γνώσεις και αυτό είναι φυσιολογικό. Επίσης, εάν αυξηθεί το κόστος παραγωγής, τότε θα γίνει και πιο ακριβό ένα προϊόν. Αυτό είναι φυσικό επακόλουθο και εδώ πρέπει και ο καταναλωτής να αναρωτηθεί αν είναι έτοιμος να πληρώσει περισσότερα χρήματα για να πάρει ένα βιολογικό ε, προϊόν. Αυτό όμως είναι δύσκολο να το κρίνω και να σας απαντήσω. Επίσης, ε, η η εισαγωγή ενός συγκεκρι... μιας συγκεκριμένης οριακής Αυτό θα αποτελέσει εμπόδιο στους ε, παραγωγούς και τους καταναλωτές ή όχι. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Φυσικά έχει πολύ, ε, πολλά πλεονεκτήματα για το περιβάλλον το να μην υπάρχουν αυτά τα κατάλοιπα, το να καταργηθούν. Τώρα, αν θα σταθεί εμπόδιο, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι μπορεί να αποτελέσει έναν κίνδυνο για πολλές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες θα έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην παραγωγή τους εάν καταργηθούν αυτές ε, οι οριακές τιμές. Πρέπει πάνω απ' όλα να λάβουμε υπόψη ε, πόσο περιθώριο έχουμε για ελιγμούς όσον αφορά τις επιδόσεις. Στη Γερμανία πάνω από 20 χρόνια διεξάγονται αναλύσεις που συγκρίνουν τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις με τις συμβατικέ. και οι αναλύσεις αυτές έχουν δείξει ότι κατά μέσο όρο οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις μπορούν να είναι κερδοφόρε. Όμως, αυτές οι αναλύσεις δείχνουν επίσης ότι περίπου 40% των βιολογικών εκμεταλλεύσεων θα ήταν πιο κερδοφόρες εάν γίνονταν συμβατικές εκμεταλλεύσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει και μεγάλο περιθώριο για ελιγμούς, ε, γιατί αυτό συνεπάγεται και επιπρόσθετο κόστος, το βιολογικό θέλω να πω. Πρέπει λοιπόν να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Τώρα, Πιστεύω πως ε, δεν έχουμε την ε, πολυτέλεια να μην κάνουμε τίποτα. Η συνθήκη της ε, Λισαβόνας πρέπει να είναι γνώμονάς μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται η βιολογική η γεωργία, να υπάρχει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο γι' αυτό και εδώ η πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα πρώτο βήμα. Βλέπω φυσικά πως επιδέχεται μεγάλες βελτιώσεις, μεγάλων βελτιώσεων, αλλά γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ. Μας καλέσατε για να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας βασισμένες στην πολυετή μας εμπειρία και ελπίζουμε αυτό να βοήθησε. Όμως πιστεύω πως μία εμπεριστατωμένη εκτίμηση επιπτώσεων χρειάζεται πολύ περισσότερες αναλύσεις και πολύ περισσότερες πληροφορίες. Εφόσον φυσικά μας ζητήθείτε κάτι τέτοιο, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο της ε, δημόσιας ακρόασης. Θα... Περάσουμε τώρα στο δεύτερο τμήμα της ε, δημόσιας ακρόασης με τρεις εμπειρογνώμονες. Παρακαλώ να λάβουν θέση στο Προεδρείο. Ελάτε παρακαλώ γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Μετά τις ε, παρεμβάσεις των τριών ε, καλεσμένων μας θα συνεχίσουμε τη συζήτηση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 σας θέλω, παρακαλώ ακριβώς λόγω της πίεσης χρόνου να περιοριστούμε στην υποβολή ερωτήσεων και όχι παρουσίασης απόψεων για να προλάβουν οι εμπειρογνώμονες να απαντήσουν. Ας αποφύγουμε λοιπόν τις δηλώσεις και τα σχόλια. Ας εστιαστούμε σε ερωτήσεις μόνο. Είναι έτοιμοι οι καλεσμένοι μας. Ο πρώτος εμπειρογνώμονάς μας για στο δεύτερο γύρο είναι ο κύριος Ετχέν Γκανιαγόν. Κύριε Τιέν Γκανιερό, είστε ο πρώτος εμπειρογνώμονας του δεύτερου τμήματος. Ε, όπως σας είπα, πίεση χρόνου υπάρχει, γι' αυτό και έχετε μόνο ένα δεκάλεπτο. Παρακαλώ κύριε Γκανιερό. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ε, γεωργός εδώ και 17 χρόνια, καλλιεργώ βιολογικό προϊόντα στο κέντρο της Γαλλίας παράγω δημητριακά, έχω αγελάζει για την παραγωγή ε, κρέατος. Λοιπόν, εκπροσωπώ τον τομέα της γεωργίας, ε, αλλά μιλάω βέβαια και για τη βιολογική καλλιέργεια, τη βιολογική γεωργία. Έχω διαφάνειες ε, που είναι αρκετά πλήρεις. Για λόγους χρονικών περιορισμών ε, μείωσα κάπως ε, της διαφάνειας όσον αφορά τη γαλλική γεωργία. Σας επέτοιμασα πολλές διαφάνειες. Βλέπετε εδώ τις, τις καμπύλες. Αύξηση της παραγωγής τα τελευταία 20 χρόνια με κατανομή, βλέπετε την κατανομή, πολύ μεγαλύτερη ποικιλομορφία στη δεξιά στήλη έχουμε τη βιολογικά προϊόντα σε σύγκριση με τη συμβατική γεωργία, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές. Ε, είναι λογικό αυτό λόγω της ποικιλομορφία που υπάρχει στην βιολογική καλλιέργεια. Όσον αφορά τι καλλιέργειε, δεν υπάρχουν μεγάλε διαφορέ. Θα καθυστερήσω κάπως αυτό το γράφημα, όπου βλέπετε μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο ιστόγραμμα είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάμεικτης παραγωγής, μίξης. Βλέπετε στον τομέα της βιολογικής παραγωγής της Γεωργία πάνω από 40% ε, των εκμεταλλεύσεων είναι μεικτές. Και εξού και το όλο πρόβλημα που αναφέρθηκε στην πρώτη συζήτηση. Βλέπουμε την αγορά, βλέπουμε πολύ κανονική αύξηση, συνεχή αύξηση της ζήτησης από πλευράς καταναλωτών η ανάπτυξη ολογική καλλιέργεια στη Γαλλία είναι αποτέλεσμα πραγματικού προγραμματισμού στη Γεωργία. Το, αριστερά το στο διάγραμμα βλέπετε στο σκούρο γαλάζιο είναι η γαλλική παραγωγή. Τα υπόλοιπα είναι εισαγωγέ. Πάνω από τα τρία τέταρτα λοιπόν τη παραγωγή βιολογικών προϊόντων που καταναλώνουν οι Γάλλοι καταναλωτέ προέρχονται από την γαλλική καλλιέργεια, από τις γαλλικές εκμεταλλεύσεις. Όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού που συζητάμε, ε, τις αρχές και το όλο πλαίσιο δεν βρήκαμε πραγματικό σχέδιο, πραγματικό πρόγραμμα που να αντιστοιχεί σε αυτή τη ζήτηση που διαπιστώνεται από πλευράς καταναλωτών. Ε, υπενθυμίστηκε από τους βουλευτές. Δεν βρήκαμε στα προ... στις αιτιολογικές ε, σκέψεις βρήκαμε μόνο τις βασικές αρχές της ε, βιολογική παραγωγή. Είναι πραγματικά σωστή νομοθεσία για ανάπτυξη τη βιολογική καλλιέργεια στην Ευρώπη. Είναι ένα ερώτημα και δεν βρήκαμε πραγματική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Όσον αφορά τι πράξη, πράξης, συμφωνούμε όλοι λίγο πολύ όσον αφορά τα κεφάλαια 2, 3 και 6 τις τεχνικές διατάξεις που αφορούν την παραγωγή, οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ σημαντικές για μας και θα πρέπει να γνωστοποιούνται σαφώς μέσω του κειμένου και όχι μέσω των κατεξισοδότης συμπράξεων όσον αφορά τις μικτές καλλιέργειες. Σε σχέση με αυτά που προανέφερα, οι μικτές καλλιέργειες στη Γαλλία είναι σημαντικές. Η κατάληψη του μεικτού χαρακτήρα των καλλιεργιών θα, θα έπεφερε περιπλοκές για την τροποποίηση και θα μειωνόταν η παραγωγική δυνατότητα στη Γαλλία. Και τα αποτελέσματα θα ήταν τα αντίθετα από την επιδιωκόμενα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραμμα δράσης, δηλαδή μείωση των προϊόντων των βιολογικών, αλλά αύξηση των εισαγωγών. Άρα η, μικτές, η εγκατάλειψη των μεικτών καλλιεργειών δεν είναι καλή ιδέα τώρα, σε αυτή τη φάση μακροπρόθεσμα μπορούμε να το κουβεντιάσουμε, εν πάση περιπτώσει όμως χρειάζεται χρόνος για κάτι τέτοιο, Όσον αφορά τα βιολογικά φυτά και τους σπόρους, χρειάζεται μεγαλύτερη παραγωγή στο βιολογικό τομέα, αλλά η χρήση των σπόρων από τους συμβατικούς σπόρους είναι κάτι που παραμένει απόλυτα αναγκαίο, ε, κυρίως ε, αν θέλουμε να έχουμε εναρμόνιση ε, των διαφόρων χωρών. Ε, που δεν, λοιπόν, η παραγωγή όταν δεν βρίσκουν σπόρους βιολογικούς πάνε σε βάση δεδομένων και προσπαθούν να βρουν την ισοδυναμία. Και το σύστημα λειτουργεί αρκετά καλά. Υπάρχει κάποια εναρμόνιση των στοιχείων. Λοιπόν, όσον αφορά τις ζωοτροφές, προτείνουμε να παραμείνουν τα όρια, αλλά να αντικατασταθούν ε, οι περιφέρειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή 90% των ζωοτροφών που πηγαίνουν στα, για, τα, για, τα βοηδή, τα τα πρόβατα, τις κατσίκες κλπ. να προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε 95% των ε, ζωοτροφών να είναι βιολογικά και να προσφύγουμε σε 50% συμβατικών συστατικών. Είναι κάτι απαραίτητο σήμερα για, αρκετές, για αρκετούς τομείς. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα όρια της ε, μόλυνσης, είναι πραγματικό θέμα αυτό, ζήτημα. Και εδώ συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να αλλάξει η φυστάμενη νομοθεσία. Υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες ε, διαφορές στην πράξη ε, και εκεί είναι που πρέπει να δημιουργήσουμε στο των καταναλωτών. Έχουμε ταξινόμηση των προϊόντων με όρια τελείως διαφορετικά και σχέδια δειγματοληψίας και ελέγχων που ποικίλουν πάρα πολύ, ακόμα και εντό ενός ε, ίδιου κρατούς μέλους. Ε, στην ε, Γαλλία οι οργανισμοί πιστοποίησης δεν έχουν το ίδιο όριο από εκμετάλλευση εκμετάλλευση όσον αφορά την ταξινόμηση και αυτό είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε και όλη αυτή η εναρμόνιση θα πρέπει να γίνει στα κράτη-μέλη, αλλά προφανώς αν μπορεί να συνοδεύεται αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή να γίνουν περισσότερα από αυτά που γίνονται σήμερα. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει. Λοιπόν, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ίσως είναι κάπως ε, πρώιμη. Ε, τούτου λεχθέντος ε, υπάρχει ανάγκη να συνεχίσουμε επεξεργασία του θέματος, το είπα και το επαναλαμβάνω και το επιβεβαιώνω θα πρέπει λοιπόν ε, να προχωρήσουμε όσον αφορά τα επόμενα σημεία. Εναρμόνιση των μεθόδων της, ε, των ερευνών όσον αφορά ε, τους ελεκτικούς φορείς, εναρμόνιση των μεθόδων έρευνα όσον αφορά ε, τα διάφορα στοιχεία που μολύνουν τα προϊόντα στα εργαστηρία θα πρέπει να υπάρξει εραρμόνιση των διαφόρων ε, πιστοποιητικών οργανισμών αν δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, να υπάρχουν διαφορετικέ δράσει όταν φτάνουμε τα όρια συναγερμού, να καθορίσουμε ακριβώ το μηχανισμό αποζημίωση επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τους ελέγχους, θα πρέπει όλες οι διατάξεις για τους ελέγχους να μπουν σε αυτό τον κανονισμό για τη βιολογική καλλιέργεια. Θα πρέπει να υπάρχει ετήσιος ελάχιστος έλεγχος κατά ε, φορέα και τεχαίοι ε, ξαφνική έλεγχη. Θα πρέπει ε, να υπάρχει δυνατότητα σε, και εκείνων που, ε, που πολύ συσκευασμένα προϊόντα να μην απαιτείται να έχει πιστοποίηση. Υπάρχουν διάφορα είδη πιστοποίηση στη Γαλλία είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, η πιστοποίηση και για τους καταναλωτές, για την ασφάλεια του καταναλωτού, αλλά και για τους παραγωγούς. Τα συστήματα πιστοποίησης είναι κάτι ε, σημαντικό για τους παραγωγούς που δέχονται το κόστος αυτού ε, και ε, πράγματι δίνει προστιθέμενη αξία. Χρειάζεται όμως έλεγχη. και αυτό διαφοροποιεί τη βιολογική καλλιέργεια από πάρα πολλά άλλα συστήματα. αντίθετα, θεωρούμε ότι σίγουρα υπάρχουν λίγα προβλήματα όσον αφορά την παραγωγή, αλλά το βασικό ε, πρόβλημα αφορά ε, τις αγωγές. Θα πρέπει οι εισαγωγές να μπουν στο πλαίσιο της συμμόρφωσης και θα πρέπει η πρόταση να συνοδεύεται από ειδικές διατάξεις για τις ε, διάφορες καλλιέργειες σε υπερπόντια εδάφη, σε περιοχές του σημερινού και και τροπικές περιοχές. Λοιπόν, ε, μετά όσον αφορά τις μεικτές καλλιέργειες και τους ελέγχους, εμείς εκπροσωπούμε τους βιολογικούς καλλιεργητές της Γαλλίας, ε, προβληματιζόμαστε από την πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πρότεινε την απαγόρευση των μεικτών καλλιεργιών παρά, και μόνο για τους καλλιεργητές, ούτε για τους διανομής, ούτε για τους μεταποιητές. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος ε, να μην συνεχιστεί, να μην επιτρέπεται η μεικτή ε, καλλιέργεια για όλους τους τομείς αλλά κυρίως για τον τομέα των, της παραγωγής. Δράτω με τις ευκαιρίες για να κλείσω με τις διαφάνειές μου καλώντας σας ε, σε μια έκθεση όσον αφορά τις βιολογικές καλλιέργειες που ε, κάθε δύο χρόνια γίνεται στη Γαλλία. Έγινε ευρωπαϊκή έκθεση, ε, λέγεται Tech and Bio. Bio. Είσαστε ευπρόσδεκτοι στη Valence για να έρθετε να δείτε τι έχουμε να παρουσιάσουμε όσον αφορά τις βιολογικές καλλιέργειες στη Γαλλία. Λοιπόν, αυτά ίσως να προχώρησα πιο γρήγορα από το χρόνο που διατέθη, όμως έτσι κερδίζουμε κάποιο χρόνο για την συζήτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκανιερό. Είστε ο πρόεδρος της ε, Agence Bio από τη Γαλλία. Θα δώσω τώρα το λόγο στην δεύτερη καλεσμένη μας, την κυρία Ισαμπέλα Ιμπερτσμπέργκερ που είναι βιοκαλλιεργήτρια και μέλος ε, της, του δικτύου νέων βιοκαλλιεργητών από την Αυστρία. Έχετε το λόγο κυρία Ιμπερτσπέργκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας ε, καλημερίσω και να σας ε, δώσω μία εικόνα του τι κάνουμε. Εμείς είμαστε μία βιολογική εκμετάλλευση κτηνοτροφική γάλακτος, βρισκόμαστε στις Άλπεις και ανήκουμε στον ε, σύνδεσμο Bank Βιολογική Αυστρία για τη Νέα Γενιά. Η βιολογική μας εκμετάλλευση λοιπόν ασχολείται με παραγωγή βιολογικού γάλακτος από αγελάδες οι οποίες βόσκουν ελεύθερα. Και είμαστε όπως είπα μια βιολογική εκμετάλλευση στην οποία ανήκει, ανήκουν βοσκότοποι και δάσος. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση και έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλους τους ε, απασχολούμενους. Τα ζώα μας βόσκουν έξω όταν ο καιρός το επιτρέπει, τουλάχιστον 120 μέρες ε, το χρόνο. Και πιστεύουμε πως ε, η τροφή την οποία λαμβάνει η αγελάδα μόνη της, όταν βοσκεί μόνη της, είναι η καλύτερη πηγή πρωτεΐνης που μπορεί να λάβει. Σύνθημά μας είναι το εάν είναι η αγελάδα καλά, είναι και ο αγρότης καλά. Το καλοκαίρι το βασικό συντηρέσιο ε, για τις αγελάδες μας είναι λιγαριά και σανό. Το χειμώνα έχουμε ε, συμπυκνωμένη ζωοτροφή την οποία δίνουμε στα ζώα μας, όμως δεν υπερβαίνει το 15%. Αυτή η... Αυτός ο τρόπος διατροφής πιστεύουμε πως είναι πάρα, ε, πάρα πολύ καλός για τα ζώα. Επίσης, Έχουμε μάθει πάρα πολλά από την εμπειρία των Γερμανών αγροτών και κτηνοτρόφων. Πιστεύουμε πως η δουλειά μας είναι κάτι που πρέπει να περιλαμβάνει πάρα πολλούς τομείς. Πιστεύουμε πως η διαβίου μάθηση είναι πάρα πολύ σημαντική για την ε, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Επίσης, ε, θα ήθελα να σας μιλήσω για τους ελέγχους. Γίνονται έλεγχοι, ξαφνικοί έλεγχοι, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στην ε, επιχείρησή μας, από ανεξάρτητες και διάφανες ε, και από ανεξάρτητους και διάφανους φορείς. Οι βιολογικοί αγρότες δεν παράγουν μόνο υψηλής ποιότητα τρόφιμα, αλλά πιστεύουμε πως συνεισφέρουν και στο περιβάλλον με μια καλύτερη ε, ποιότητα τροφίμων, με αύξηση της βιοπικιλότητας και με ένα ε, τοπίο το οποίο είναι και αισθητικά όμορφο και προς, αυξάνει τον τουρισμό επίσης. Πιστεύουμε πως η πρόταση για τις οριακές τιμές ε, καταλήπων είναι λάθος. Εμείς ε, πιστεύουμε σε μια κατάργηση των οριακών τιμών καταλήπων, διότι είναι ο πιο δίκαιος ε, τρόπος παραγωγής. Επίσης πιστεύουμε πως ε, πρέπει να ενισχυθεί η διαδικασία ελέγχου και να ενισχυθούν και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ε, μιας βιολογικής εκμετάλλευσης. Η ξαφνική επιτόπη έλεγχη πιστεύουμε πως είναι μια σωστή και μακροπρόθεσμη, μακροπρόθεσμα εφικτή μέθοδος. Η η εκμετάλλευσή μας βρίσκεται στο Ζάλσπουργκ της Αυστρίας και είμαστε η πρώτη σε παραγωγή βιολογικών προϊόντων περιφέρεια της Ευρώπης. Το 50% της παραγωγής μας είναι βιολογική παραγωγή και βρισκόμαστε στην πρώτη θέση των ε, παραγωγών βιολογικών προϊόντων. Το γάλα που παράγουμε είναι βιολογικό και μόνο 3% του γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή προέρχεται από βιολογικές πηγές με τον τρόπο ε, που έχουμε τα, ε, που διαχειριζόμαστε τα ζώα μας. Χωρίς συντηρητικά και χωρίς περιττή επεξεργασία. Αυξάνεται επίσης και η ζήτηση για τα βιολογικά προϊόντα και για το βιολογικό ε, γάλα. Και πιστεύω πως ε, τα χρονοδιαγράμματα δεν είναι τα επιθυμητά. Όπως σας είπα, αυξάνεται ένα και περισσότερο η ζήτηση σε βιολογικά προϊόντα, σε βιολογικό γάλα. Και πιστεύουμε πως οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις που ε, περιλαμβάνουν και δασικές εκτάσεις και διάφορες ε, καλλιέργειες και εκτινοτροφικές ε, μονάδες είναι ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης όχι μόνο των ίδιων των προϊόντων αλλά και του περιβάλλοντος. Χρειάζεται επίσης και αυξημένη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των καταναλωτών, διότι βλέπουμε πως υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των καταναλωτών και χρειάζεται λοιπόν να δοθεί προσοχή σε αυτό. Επίσης χρειάζεται και αύξηση της ε, δυνατότητας δικτύωσης των ε, αγροτών, ιδιαίτερα των ε, νεότερων αγροτών. Από το 2015 και μετά ο σύνδεσμός μας για τους νέους ε, βιολογικούς αγρότες στην Αυστρία θα έχει συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένες ε, ποσοστώσεις και θα μπορέσει να δεχτεί περισσότερους, περισσότερα μέλη. Τώρα, το κίνητρο που έχουμε. Το κίνητρο που έχουμε είναι η βιολογική γεωργία. Η βιολογική γεωργία είναι ε, βιώσιμη, αϊφόρος και πιστεύουμε πως ε, φροντίζει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη για την επόμενη γενιά, όχι μόνο τη δική μου αλλά και τη γενιά των παιδιών μου. Τα βιολογικά προϊόντα φυσικά αποτελούν μια μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά και, και προϋποθέτουν επίσης μεγαλύτερη κατανόηση της φύσης και του ζώου. Αλλά αυτό είναι συνάμα και το ευχάριστο. Ο κανονισμός για τα βιολογικά προϊόντα αποτελεί μια πάρα πολύ καλή βάση για την ε, δουλειά μας και η αλλαγή, η τροποποίηση σε σημαντικό βαθμό αυτού του κανονισμού θα επηρεάσει πάρα πολύ την ε, δική μας ε, τη δική μας δουλειά, τη δική μας ζωή. Πρέπει να δείτε τα πράγματα από τη δική μας επίσης σκοπιά. Σας μίλησα ήδη για το γιατί διαφωνώ με, την, με τις ε, οριακές τιμές καταλήπων. Και όσον αφορά τις μικτές εκμεταλλεύσεις, θα ήθελα να πω ότι εμείς έχουμε συγκεκριμένες προδιαγραφές στο, στο οργανόγραμμά μας, στον τρόπο λειτουργίας μας, και πιστεύουμε πως ε, καλό θα ήταν να ε, καταργηθούν οι μεικτές εκμεταλλεύσεις και να μετατραπούν σε βιολογικές. Φυσικά αυτό χρειάζεται μια σταδιακή αλλαγή και πιστεύουμε πως ε, οι λύσεις που έχουν προταθεί από τον κανονισμό δεν είναι οι κατάλληλες. Διότι αυξάνουν το κόστος της ε, μεταβολής και θα δημιουργήσουν ενδεχομένω φραγμούς στη διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Επίσης, τι περιμένω από την εφαρμογή του κανονισμού εάν αυτός εφαρμοστεί όπως είναι. Περιμένω μία μείωση της παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Γι' αυτό λοιπόν και είναι αναγκαία μία τροποποίηση, είτε τροποποίηση όσον αφορά τις ε, ζωοτροφές, είτε τροποποίηση όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά και τους ελέγχους. Θεωρώ ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής είναι πάρα πολύ επικίνδυνη πιθανά, διότι θέτει σε κίνδυνο τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις, δεν τις ε, ενισχύει, αλλά απειλείται η ίδια τους η ύπαρξη, διότι πάρα πολλοί αγρότες δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν βιολογικά θα ήθελα να σας κάνω μία έκκληση, να μην μας ξεχνάτε, διότι εμείς προσπαθούμε όσοι η νέα γενιά αγροτών να χτίσουμε το μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε έναν εφαρμόσιμο και λογικό κανονισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η τελευταία μας καλεσμένη, κυρία Ελία Ροντρίγες Άλβαρες που είναι βιοκαλλιεργήτρια και εκπρόσωπος της Αγροτικής Ένωσης της Γαλλικίας. Παρακαλούμε κυρία Άλβαρες, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Δεν συνηθίζω να μιλάω σε τόσο μεγάλη ομιγύρη. Γι' αυτό σας ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη για την αμηχανία μου. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη χρειάζεται βιολογικές καλλιέργειες και βιολογικά προϊόντα. Και καλό θα ήταν να μειώσουμε τις συμβατικές καλλιέργειες και να τονώσουμε και να ενισχύσουμε τις βιολογικές. Μια βιολογική καλλιέργεια, μια βιολογική γεωργική εκμετάλλευση όπως ξέρετε, βελτιώνει την ποιότητα ζωής και του γεωργού, αλλά ταυτόχρονα βελτιώνει το περιβάλλον, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, κάτι που είναι ιδιαίτερο σημαντικό. και ταυτόχρονα φέρνει τον κόσμο στην Ήπεθρο ε, με νέους ή λιγότερο νέους γεωργούς όπως υποφαινομένοι. Και επίσης δημιουργεί τοπίο γιατί η ύπεθρός μας απεριμόνεται. Υπάρχει μια στιφιλία, μια έξοδος από τις αγροτικές ζώνες και από την η ηπεθρος Επίσης δίνεται μια στιφιλια μια εξοδος απο τις αγροτικες ζωνες και απο την ηπεθρο επισης δινεται μια εμφαση στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις και οι μικρές εκμεταλλεύσεις ε, πεθαίνουν. Στη Γαλλική έχουμε κάθε καλοκαίρι πυρκαγιές, οπότε η ύπεθρός μας ερημώνεται. Όταν είχαμε γεωργούς στην ύπεθρο, είχαμε πολύ λιγότερες πυρκαγιές ή σχεδόν καθόλου, ή τις θέταμε πολύ εύκολα υπό έλεγχο. Τώρα, επειδή οι γεωργοί έχουν εγκαταλείψει την ύπεθρο, οι πυρκαγιές αυξάνονται. Ασχολούμαι με την ε, βιολογική καλλιέργεια εδώ και πολλά χρόνια. Είναι αυτό το το βιοποριστικό μου επάγγελμα και θεωρώ ότι η βιολογική γεωργία θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό θα πρέπει να μειώσουμε την ε, συμβατική γεωργία. Δεν είναι θέμα να έχουμε περισσότερους κανονισμούς ή λιγότερους κανονισμούς. Το θέμα είναι ε, μακροπρόθεσμα να διαλέξουμε μία αηφόρο, βιώσιμη γεωργία, για να μπορούν και τα παιδιά μας και οι απογονοί μας να καλλιεργούν τα ίδια εδάφη και τα ίδια χωράφια που καλλιεργούμε εμείς σήμερα γιατί με το ρυθμό που προχωρούμε και με την ποσότητα ζυζανιοκτώνων και φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούμε στη γεωργία, η γεωργία δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Οπότε χρειαζόμαστε, δεν ξέρω αν το πω βοήθεια, γιατί μιλήσαμε για τους σπόρους. Εγώ χρησιμοποιώ κατά το ίμιση τους δικούς μου σπόρους. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να αναπαράγουμε αυτούς τους σπόρους. Δεν ξέρω, αν χρειάζονται πιστοποίηση, ποιο θα το κάνει. Εγώ δεν μπορώ να κάνω την πιστοποίηση των δικών μου σπόρων, άρα χάνουμε αναπαραγωγικό υλικό, χάνουμε γενετικό υλικό, πολλαπλασιαστικό υλικό των φυτών. Οπότε στον κανονισμό θα πρέπει να προβλέψουμε τη δυνατότητα ανταλλαγή σπόρων μεταξύ των γεωργών. Υπό τον όρο ότι ε, είναι βιολογικές όλες αυτές οι καλλιέργειες, γίνεται ανταλλαγή σπόρων μεταξύ των βιοκαλλιεργητών και για βιολογικούς σπόρους. Δυστυχώς στην ε, Ισπανία υστερούμε στην έρευνα. Εγώ για να βρω οικολογικούς, βιολογικούς, πιστοποιημένους σπόρους πρέπει να τους αγοράσω από την Αυστρία ή από τη Γαλλία ή από τη Γερμανία. Στην πατρίδα μου την Ισπανία δεν έχουμε επιχειρήσεις ε, που παράγουν τέτοιους σπόρους ή που τους κρατάνε. Μπορεί να έχουμε ελάχιστες ε, ε, επιχειρήσεις που ασχολούνται με το θέμα αυτό, αλλά είναι πολύ μικρές οι δόσεις, πανάκριβες και δεν ξέρουμε αν ανταποκρίνονται στις ε, γεωγραφικές ε, και δαφολογικές συνθήκες της Ισπανίας. Γιατί δεν σημαίνει ότι ένας πόρος που ευδοκιμεί στην Αυστρία θα ευδοκιμήσει και στην Ισπανία. Οπότε χρειαζόμαστε έρευνα για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τους πιστοποιημένους πόρους στις εδαφολογικές και κλιματικές ιδιαιτερότητες της Ισπανίας και της κάθε περιφέρειας της Ισπανίας και χρειαζόμαστε περισσότερη βοήθεια και στήριξη για να αυξήσουμε την παραγωγή μας. Εγώ δεν λαμβάνω τίποτα, καμία υποστήριξη, καμία βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η βοήθεια δίνεται αναέκταση και για τις, ε, μικρές, για τις μικρές εκτάσεις ε, δεν υπάρχει καμία τέτοια βοήθεια. Η δική μου γεωργική έκταση είναι πολύ μικρή, οπότε ούτε καν μπαίνω στον κόπο να ζητήσω επιδότηση. Γιατί θα ξοδέψω πολύ περισσότερα για να υποβάλω την αίτηση από ό,τι θα είναι το ποσό της επιχορήγησης. Οπότε στην Ισπανία οι μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις λαμβάνουν τις ε, ενισχύσεις. Γιατί η ενίσχυση πια γίνεται με βάση την γεωργική έκταση και όχι με βάση την παραγωγή. Άρα οι μικρές εκτάσεις και οι μικροκαλλιεργητές πλήττονται, βρίσκονται σε δυσμενή θέση. Η κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων αυξάνεται, όπως είπαμε, με σταθερούς ρυθμούς. Και γι' αυτό πρέπει να αυξήσουμε και την βιολογική παραγωγή για να καλύψουμε τη ζήτηση σε βιολογικά προϊόντα. Και δεν μιλώ, εγώ δεν θέλω μία ελιτιστική παραγωγή, ούτε θέλω να παράγουμε βιολογικά προϊόντα μόνο για τους ευπόρους, για αυτούς που έχουν την πολυτέλεια να αγοράζουν τέτοια προϊόντα. Θέλουμε να είναι βιολογικά τα, τα προϊόντα σε όλο... για όλο τον κόσμο. Δεν με ενδιαφέρει να έρχονται μόνο οι εύποροι που έχουν υψηλή αγοραστική δύναμη και να αγοράζουν βιολογικά προϊόντα. Και οι υπόλοιποι δηλαδή ο απλός κόσμος τι θα τρώει. Δεν θα έχει πρόσβαση στα βιολογικά προϊόντα επειδή είναι ακριβά. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να στηρίξουν την ε, βιολογική γεωργία για να καταστήσουν τα βιολογικά προϊόντα προσιτά σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και όχι μόνο σε μία ελίτ προνομιούχα που έχει υψηλή αγοραστική δύναμη. Επίσης, αν έχουμε έναν άκαμπτο κανονισμό, θα ευνοηθούν οι χώρες ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πιο χαλαρούς ε, κανονισμούς. Οπότε ξεχάστε την ε, ανταγωνιστικότητά μας θα μπορέσουμε να συναγωνιστούμε άλλες χώρες που εξαιτία χαλαρών ε, νομοθεσιών θα έχουν πιο φθηνή παραγωγή. Επίσης, ε, τα μέτρα θα πρέπει να ισχύουν για όλους. Οι αυστηρές προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωση θα πρέπει να ισχύουν και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Αλλιώ οι Ευρωπαίοι παραγωγοί θα τεθούν σε δυσμενή θέση. Επίση, τα μη βιολογικά προϊόντα δεν έχουν τέτοιε επιβαρύνσεις εμείς οι βιοκαλλιεργητές πρέπει να πληρώνουμε για την πιστοποίηση. Και ποιος πληρώνει την πιστοποίηση, η ίδια παραγωγή, οι καλλιεργητές. Ενώ θα πρέπει τα θεσμικά όργανα, κατά τη γνώμη μου, να πληρώνουν τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων. Όχι η γεωργία από την τσέπη τους, γιατί εγώ πληρώνω στο Συμβούλιο το Ρυθμιστικό της Γαλλικίας ένα ποσό για να πιστοποιήσει ότι η παραγωγή μου είναι βιολογική. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι άδικο να πληρώνουν από την τσέπη τους οι γεωργοί την πιστοποίηση των προϊόντων τους. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, για να απαντήσω σε κάποιες απορίες. Το όριο των καταλήπων. Αν τα κατάλοιπα είναι της ίδιας της αγροτικής εκμετάλλευσης και γι' αυτά φταίει ο Γεωργός, κανονικά θα πρέπει να είναι μηδενικά τα κατάλοιπα αλλά δυστυχώς ε, υφιστάμεθα επιμόλυνση έξωθεν. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον αέρα που έχει ατμοσφαιρική ρήπανση. Δεν φταίμε εμείς για την ατμοσφαιρική ρήπανση, ρήπανση συγγνώμη. δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα του αέρα και το νερό μπορεί να είναι μολυσμένο. Δεν φταίμε εμείς όμως αν το νερό που φτάνει στην εκμετάλλευσή μας δεν είναι καθαρό. Κατά τη γνώμη μου όντως σε μια βιολογική εκμετάλλευση τα κατάλοιπα θα πρέπει να είναι μηδενικά. Αλλά δυστυχώς ε, ζούμε μέσα σε ένα μολυσμένο περιβάλλον. Επίσης, αν ο γείτονα μου είναι συμβατικός Γιώργος, τι να κάνω, να πάω να τον καταγγείλω επειδή μολύνει τη δική μου βιολογική παραγωγή. Τι φταίει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπο δεν έχει επιλέξει το βιολογικό μοντέλο παραγωγής, αλλά δικαιούται να παράγει και να ζήσει. Προτιμώ να κλείσω τη δική μου βιολογική παραγωγή παρά να καταγγείλω το γειτονά μου και να τον εξωθήσω στην ανεργία. Οπότε είναι αναπόφευκτη από τη στιγμή που γετινιάζουν συμβατικές με μη συμβατικές ή βιολογικές καλλιέργειες να υπάρχει κάποια επιμόλυνση. Η έβδομη ερώτηση, που είναι δύσκολο να απαντήσω. Πιστεύω ότι ο κανονισμός θα πρέπει να είναι σοβαρός, που θα επιτρέπει την παραγωγή υγιεινών προϊόντων, που δεν θα ρηπαίνουν το περιβάλλον, είναι εύλογος αυτός ο στόχος, αλλά δεν ξέρω αν είναι η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει ένα τέτοιο κανονισμό. Δεν μπορώ να δώσω εγώ μια τέτοια απάντηση. Πάντως, ε, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται εκτενή συζήτηση, διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους, γιατί εμείς ε, είμαστε ένα τμήμα της παραγωγής και ένα τμήμα της ζωής. Αυτά. Ακούσαμε με ιδιαίτερη χαρά τους εμπειρογνώμονές μας. Πραγματικά ε, διαλευκάναμε πολλά σημεία και επιπλέον ευχαριστώ θερμά τους εμπειρογνώμονες γιατί τήρησαν όλοι το χρόνο που είχαν και θα πρέπει να τους μιμηθούμε και εμείς. Μην ξεχνάτε ότι στις 12 παρατέταρτο πρέπει να κλείσουμε τη συνεδρίασή μας γιατί ακολουθεί η συνεδρίαση των συντονιστών. Οπότε έχουμε ελάχιστο χρόνο, ουσιαστικά 20 λεπτά. Ένα λεπτό στον καθένα θα δώσω αυτή τη φορά. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρατηρήσεις που έκαναν όλοι οι συγητές. Πιστεύω να καταφέρουμε να βρούμε ένα σωστό πλαίσιο έτσι ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται ο τομέας της βιολογικής καλλιέργειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε τους βιολογικούς καλλιεργητές, τους βιολογικούς αργρότες, αλλά επίσης και να μην ξεχνάμε τους καταναλωτές, διότι τα προϊόντα... Ε, καταλήγουν σε εκείνους. Εκείνοι είναι οι τελικοί χρήστες των βιολογικών προϊόντων. Πρέπει φυσικά να σκεφτούμε τους ε, καταναλωτές, να σκεφτούν ε, εκείνους που, χρειά, που θέλουν να αγοράσουν βιολογικό κρασί, ε, τυρί, γάλα. Πιστεύω πως είναι μία... είναι ένας ε, χώρος στον οποίο ε, ενδεχομένω να υπάρξει απάτη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όντως να καταργηθούν τα, ε, οι τιμές κατά καταλήπων. Θεωρώ πως ακόμα και αν δεν είναι λάθος του καλλιεργητή, του παραγωγού, σε περίπτωση που υπάρχουν κατάλοιπα, δεν θα πρέπει αυτά τα προϊόντα να θεωρούνται βιολογικά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την τελευταία μας καλεσμένη για την ε, ομιλία της, γιατί όπως είπε ήταν η παρθενική της ομιλία σε ευρύ κοινό. Θα ήθελα πάντως να τη συγχαρώ γιατί ήταν ε, πολύ καλή παρά την ε, απειρία της. Είναι σημαντικό αυτό που είπατε για τους διαφοροποιημένους κανόνες. Επίσης σημαντικό είναι το θέμα των μεικτών εκμεταλλεύσεων, όπου συνυπάρχει συμβατική και βιολογική γεωργία. Σε πολλές χώρες έχουμε κατακαιρματισμένες εκμεταλλεύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε σε όλους τους γεωργούς να βγάζουν το ψωμί τους. Γιατί αν απαγορεύσουμε τις μεικτές καλλιέργειες θα είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσουν πολύ μικροκαλλιεργητές. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να εξασφαλίσουμε την επιβίωση των μεικτών καλλιεργειών. Κύριος Μπονάνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω ότι το 2021 είναι πολύ μακριά. Πρέπει να κινηθούμε πιο ε, γρήγορα. Δεν, είμαι υπέρ των καταναλωτών. Δεν υπερασπίζομαι τις πολυεθνικές. Είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τους μικρούς εκείνους που παράγουν με έναν τρόπο πιο σωστό. Πολύ συχνά αισθάνθηκα ότι στην Αυστρία κάνουν ένα χρόνο το, ε, μία έναν έλεγχο το χρόνο και το θεωρούν καινοτομία. Ε, λοιπόν, ε, κάνουν τον έλεγχο μόνο το Φεβρουάριο και δεν κάνουν άλλον. Πρέπει να είναι περισσότεροι έλεγχοι το χρόνο. Διαφορετικά πάνε όλα καλά και τελικά την πληρώνει ο καταναλωτής γιατί δεν βάζουμε τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων. Ένας καταναλωτής θέλει να ξέρει από πού φτάνει το εμπόρευμα, αν υπάρχουν πραγματικά οι έλεγχοι. Και τέλος, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, πιστεύω ότι στο κάτω-κάτω αν κάποιος αγοράζει βιολογικά προϊόντα και αγοράζει πληρώντας κάτι παραπάνω, θέλει να έχει ένα υγιές προϊόν. Εάν λοιπόν θέλει να έχει ένα υγιές προϊόν και πληρώνει παραπάνω, είναι δίκαιο να υπάρχουν λιγότερα λόγια, περισσότερη έλεγχη και μια παραγωγή προς όφελος του καταναλωτού. Ευχαριστώ κύριο Καλημέρα. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες. Ήταν έξοχες οι παρουσιάσεις τους. Είχα κάποιες ερωτήσεις ε, όσον αφορά την πρώτη εμπειρογνώμονα, είχα, μία, είχα τρεις ερωτήσεις, αλλά θα θέσω μόνο μία. Και αν οι εμπειρογνώμονες από το πρώτο μέρος της ε, ακροάσεως ε, είναι παρόντες, ίσως να μπορούν να απαντήσουν. Στην παράγραφο 61 και 62 της προτάσεως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα σύστημα ομαδικής πιστοποίησης παραγωγών για να μειωθεί το διοικητικό άχθος και οι δαπάνες. Ταυτόχρονα αναφέρεται ότι μια ομάδα επιχειρηματιών είναι μια ομάδα που κάθε επιχειρηματίας είναι ένας αγρότης, έχει μια εκμετάλλευση που δεν είναι μεγαλύτερη από 5 εκτάρια γεωργικής γης και ανήκουν στην παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών ε, και μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στη μεταποίηση των προϊόντων αυτών. Σημαίνει ότι αυτοί που θέλουν να μπουν σε αυτούς τους τομείς πρέπει να πληρούν αυτά τα παιδιτικά κριτήρια και βοηθούν αυτά τα κριτήρια. Αν παραμείνει ορισμός, σημαίνει ότι ομαδικές πιστοποίησεις απαιτούν από τον κάθε παραγωγό επίσης να συμμετάσχει στη μεταποίηση των προϊόντων. Έχετε κάποιο σχόλιο όσον αφορά αυτό. Ευχαριστώ κύριε Χάζεκαμπ. Eh, Σας ευχαριστώ. Θερμά ευχαριστώ στους καλεσμένους μας, γιατί πραγματικά τα λόγια τους ε, ε, με ενέμπνευσαν, ε, μου δίνουν εμπιστοσύνη, αλλά μου δημιουργούν και ελπίδες. Και φυσικά θέλουμε να έχουμε ζώα ελευθέρας βοσκής, να μπορούν να βγαίνουν στα λιβάδια και να βόσκουν χλωροχόρτο. Τι γίνεται όμως με κάποιες πρακτικές κακομεταχείρισης ε, ζώων. Επίσης, τα κατάλοιπα. Η βιοκαλλιεργήτρια από την ε, Ισπανία μας είπε ότι έχει πρόβλημα με τις γειτονικές καλλιέργειες που είναι συμβατικές. Ίσως θα πρέπει και στην παραδοσιακή γεωργία να μειώσουμε τη χρήση κάποιων ζενιοκτώνων και φυτοφαρμάκων για να μην επιμολύνει τόσο τη βιολογική γεωργία. Ο κύριος Ζουλόχ. Ευχαριστώ να προσθέσω, να προσθέσω. Πιστεύω ότι εντελώς βιολογική γεωργία είναι προς επιδίωξη στόχος. Για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε έναν κανονισμό που να μην είναι όμως πολύ περιοριστικός, συνεπώς να πετυχαίνει και πετυχαίνει έτσι το αντίθετο αποτέλεσμα. Σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τα διάφορα όρια τα οποία θα θεσπίσουμε εντός του κανονισμού. Είναι μια συζήτηση που θα μπορούσε να ανοίξει επίσης και όσον αφορά τα κατάλοιπα. Διότι όταν μιλάμε για βιολογικά προϊόντα δεν, χρειάζεται να, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια διαδικασία Οπότε ήδη θα πρέπει να προσέξουμε και τη διαδικασία. Είναι σημαντικό αυτό. Και το κατάλοιπο μπορεί να τεθεί σαν δευτερεύον ζήτημα. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Μια ερώτηση προς τους εμπειρογνώμονες. Θεωρώντας ότι το θέμα των μεικτών ε, εκμεταλλεύσεων είναι πάρα πολύ προβληματικό, κατά την άποψή σας, από την εμπειρία σας, ποιος είναι ο ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ούτως ώστε να μπορεί να μετατραπεί μια επιχείρηση από συμβατική εντελώς να γίνει βιολογική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μποβέ. Καλημέρα, πολύ γρήγορα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στην αρχή την όλη συζήτηση για ένα νέο κείμενο. Ε, αυτό σίγουρα λόγω των απατών που διαπιστώθηκαν στην αγορά των εισαγωγών και από εκεί ξεκίνησε το πράγμα. Γιατί λοιπόν θέλουμε εμείς να ετοιμάσουμε ένα γενικό κείμενο όταν το θέμα προς διευθέτηση είναι το θέμα της απάτης όσον αφορά τα ψευδοβιολογικά προϊόντα. Το σκάνδαλο που ξέσπασε στην Ιταλία πέρσι ήταν ένα σκάνδαλο απίθανο α, λοιπόν πάρα πολύ των 30 τόνι σόγια από διάφορε χώρε και αραβώση του που δεν ήταν βιολογικά προϊόντα από τέτοιες χώρε. Όλα αυτά που καλύφθηκαν από οργανισμού πιστοποίηση ε, και ήταν ένα σκάνδαλο, πλήρε σκάνδαλο και αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Εάν η εμπιστοσύνη του καταναλωτού ε, ανατιναχθεί διότι γίνονται εισαγωγές ψεύδο βιολογικών προϊόντων θα έχουμε ένα βασικό πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ δεν θα ήθελα σε αυτό το κείμενο και το ζητώ του εμπειρογνώμου άλλωστε να μα πούν ποια είναι η άποψή του. Δεν θα ήθελα λέγω στο κείμενο να, να είναι γενικό. Μήπω θα έπρεπε να θέσουμε το στόχο αυτό, συμφωνεί η Επιτροπή Γεωργία. Το θέμα είναι η πιστοποίηση, το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο είναι η έλεγχη. Και το τρίτο πρόβλημα που ετέθη, και σταματώ εδώ, ήταν και το θέμα ε, της ρήπανσης των καταλήπων. Εάν μολυνθεί ένας καλλιεργητής και παραχθεί ένα προϊόν και χάσει την ταξινόμηση ε, λόγω της μόλυνσης, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο. Ευχαριστώ κύριε Σοροπέ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω πως είμαι κάπως απογοητευμένος από την τοποθέτηση των εμπειρογνωμόνων σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Επιτροπής και φυσικά θέλουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, πιο ασφαλή βιολογικά προϊόντα, γιατί οι καταναλωτές έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα προϊόντα αυτά. Θα ήθελα να ρωτήσω τους εμπειρογνώμονές μας, λοιπόν, αυτά τα βιολογικά προϊόντα. Μπορούν να φτάσουν εγκαίρως στους καταναλωτές, μπορούν να φτάσουν χωρίς να έχουν αναμειχθεί με συμβατικά προϊόντα και ποιος είναι ο προσανατολισμός σας για το μέλλον όσον αφορά τους ε, κανόνες και τι θεωρείτε πως είναι πρακτικό και εφικτό. Ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις ε, για τις εξαιρέσεις των κανόνα. Πιστεύω πως ε, η εξαίρεση για τους σπόρους είναι απόλυτα κατανοητή, διότι πάρα ε, πολύ χρειάζονται Αυτού ε, του ε, βιολογικούς πόρους, όταν όμως δεν υπάρχουν πρέπει να καταφύγουν στους συμβατικούς και είναι, είναι κάπως ε, δύσκολο επίσης να εφαρμοστούν όλοι οι κανόνες της σε μικρές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις μικρές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να αλλάξουν οι εγκαταστάσεις στάβλησης των ζώων και τα λοιπά. Και ο κανονισμός ακούγεται πάρα πολύ ε, ρομαντικός, αλλά όμως πιστεύω πως είναι δύσκολο εφαρμόσιμο στην πράξη. Θα ήθελα όμως ε, να ρωτήσω όσον αφορά την, ε, μετα, την μετάβαση μιας εκμετάλλευσης, την αλλαγή, την αλλαγή σε βιολογική, τι γίνεται με, την, μετάβαση, με την μεταφορά των προϊόντων. Και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις, ε, ε, τα ανάμεικτα προϊόντα, βιολογικά και συμβατικά. Έχουμε τέσσερις ακόμη ομιλητές. Κύριε Φεράν, για ένα λεπτό, γιατί δεν μιλήσατε προηγουμένως. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσες ε, οι παρεμβάσει Όλοι είμαστε υπέρ τη ενθάρρυνσης και τη προώθησης τη βιολογική γεωργία. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε. Αλλά προσοχή. Ακούσαμε και επαγγελματίε και ευρωβουλευτέ. μην ξεχνάτε ότι έχουμε και εισαγόμενα προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, μεταλλαγμένα, ορμόνες και ούτω καθεξής. Οπότε εμείς έχουμε ε, υψηλέ προδιαγραφέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα υποστούμε τι συνέπειε ε, των ε, συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών που έχουμε συνάψει με τρίτε χώρε. Ευχαριστώ. Γκυό, Αγγιλέρα και Κιώστιγκερ. Μήπως θα μπορούσατε να παρατηθείτε, έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις ή να περάσουμε στους εμπειρογνώμονες. Άντε μισό λεπτό. Άγνιου στην Κεραγγιλέρα. Μισό λεπτό, κύριο Άγνιο. Κύριο Γκυγιώμα, άκουσα εμένα, εννοούσατε. Αγνιού. Μάλιστα, ωραία. Τις λίγες ερωτήσεις να απευθύνω προς την κυρία Χούμπεσμπεργκα. Είπατε ότι είχατε 500 αγελάδες παραγωγής γάλακτος σε 150 εκτάρια. Έτσι κατάλαβα κουνάτε το κεφάλι σας. Μου φάνηκε τελείως παράλογο. Σας παρακαλώ, μπορείτε να απορρίψετε ή να επιβεβαιώσετε μια φήμη. Μου είπαν ότι οι καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το glyphosate στην Αυστρία, μια ουσία και θέλετε πιο περισσότερη βιολογική καλλιέργεια. Αυτό δεν θα έπρεπε να, να κατευθύνεται από τους καταναλωτές περισσότερο. Διότι αν έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή από τη ζήτηση τελικά θα έχουμε πλεόνασμα βιολογικών προϊόντων και θα χάσει τη θέση που έχει. Σένερα. Κυρία Σένερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεδομένου ότι η βιολογική γεωργία δεν ε, παράγει απλώς υγιεινά προϊόντα, αλλά έχει και άλλες ε, και άλλα ωφέλη, μήπως θα πρέπει να προωθήσουμε πέραν της βιολογικής γεωργίας και την τόπια παραγωγή και την παραγωγή σε, και κατανάλωση κοντά στο χώρο παραγωγής. Κυρία Κάστιγκερ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Ροντρίγκες, μας είπατε ότι ειδικά για τις μικρές εκμεταλλεύσεις υπάρχουν ελάχιστες ευκαιρίες για να γίνει κάτι. Είμαι αυστριακή και πραγματικά πιστεύω πως ιδιαίτερα οι μικρές εκμεταλλεύσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες και ε, μεγάλο δύναμικο. Και μας είπατε ότι χρειάζεται περισσότερη στήριξη. Εσείς θεωρείτε πως η στήριξη είναι οικονομικής φύσης, ε, η στήριξη που χρειάζεται ή θεωρείτε πως ε, τα προϊόντα πρέπει να έχουν υψηλότερες τιμές στην αγορά. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγο και πάλι στου εμπειρογνώμονέ μα ε, για ένα δίλεπτο καθένα, παρακαλώ. Ο κύριο ε, Γκανιερό ή η κυρία Ιβερτσμπέργκερ. Θα αρχίσω. Θα ήθελα να διορθώσω λοιπόν τα νούμερα. Εμεί έχουμε 80 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και σε 105 εκτάρια. Ο μέσος όρος στην Αυστρία είναι 16 αγελάδες, 18 αγελάδες, με συγχωρείτε. Τώρα μας ρωτήσατε για την πρόσβαση. Στην Αυστρία σε γενικές γραμμές έχουμε υψηλότερα υψηλότερε προδιαγραφέ, αυστηρότερε προδιαγραφέ από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό συμβαίνει και επειδή έχουμε πιο ε, μακρόχρονη βιολογική παράδοση, αλλά και επειδή είμαστε ε, περισσότερο αγροτική χώρα. Στην Αυστρία θεωρούμε πως οι ενισχύσεις για την ε, βιολογική γεωργία είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ε, βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, ωστόσο προσπαθούμε και από μόνοι μας να είμαστε δημιουργικοί και να ε, αυξήσουμε τις δυνατότητές μας. Τώρα, όσον αφορά την πρόσβαση σε δυνατότητες αλλαγή μιας εκμετάλλευσης σε βιολογική, προσπαθούμε και εμείς να συνεργαστούμε με τις άλλες χώρες όσο το δυνατόν περισσότερο. Τώρα, ε, <clears throat> ρωτήσατε πότε είναι ε, η κατάλληλη στιγμή, ποιο είναι το κατάλληλο χρονικό διάστημα για να αλλάξει μια εκμετάλλευση και να γίνει καθαρά βιολογική. Πιστεύω πως το πιο σημαντικό εδώ είναι ε, να δούμε ότι η κατάλληλη στιγμή είναι όταν η αγορά καταφέρει να μας κάνει να μπορούμε να ζήσουμε από τα βιολογικά, βιολογικά μας προϊόντα. Αυτή θα είναι η κατάλληλη στιγμή της ε, ολικής αλλαγής σε βιολογική εκμετάλλευση. Euh, Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις, πολύ ενδιαφέρουσες ε, ακούστηκαν. Θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικός όσον αφορά τις μικτές εκμεταλλεύσεις. Προφανώς δεν θέμα διαρκείας ή περίοδου που τίθεται στη Γαλλία αποτελεί ένα στόχο να συνοδεύουμε τις εκμεταλλεύσεις να πάνε προς 100% βιολογικές καλλιέργειες. Υπάρχουν όμως και κάποιες τεχνικές προδιαγραφές για την παραγωγή διάθεση στην αγορά που απαγορεύουν στους παραγωγούς να έχουν όλη την εκμετάλλευσή τους στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Ένα παράδειγμα έθεσα τη ε, μελισσοκομεία. Κάποιος που παράγει μέλι αν η περιοχή που έχει δεν μπορεί να πιστοποιηθεί από τον έλεγχο, αν είναι κοντά σε ένα εργοστάσιο παραδείγματο χάρη, δεν θα μπορέσει να πιστοποιηθεί ότι παράγει βιολογικά προϊόντα. Δεν είναι λόγω τη δική του θέληση που παραμένει μεικτή καλλιέργεια γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Στη Γαλλία έχουμε και άλλε παραγωγέ όπω τα ζαχαρότευτλα, όπου υπάρχουν πολύ λίγοι ε, που χρησιμοποιούν αυτά τα βιολογικά ζαχαρότευτλα για τη βιομηχανία. Ίσως άλλες χώρες να έχουν προχωρήσει περισσότερο. Στη Γαλλία ένας παραγωγός που θέλει να περάσει τη βιολογική καλλιέργεια δεν μπορεί να θέσει στο εμπόριο τα βιολογικά του ζαχαρότευτα οπότε είναι υποχρεωμένος αν θέλει να προχωρήσει, να εγκαταλείψει αυτή την παραγωγή, ενώ ε, ίσως θα μπορούσε να είναι πιο κερδοφόρα της εκμετάλλευσης. Είναι αρκετά ευαίσθητη λοιπόν η επιλογή. Τώρα για την ευημερία των ζώων τέθηκε ένα ερώτημα. Ε, ε, κινούμεθα πιο γενικά, είναι πιο ευρύ το θέμα, το συζητάει η κοινωνία, πιο πέρα από τον κανονισμό, είναι δύσκολο το θέμα, διότι ακόμα και τη βιολογική παραγωγή υπάρχουν πρακτικές που ακολουθούνται που θεωρούμε ότι επιβάλλονται συναρτήσει της, ε, ε, ε, της αγοράς όπως ο ευνοχισμός των σενικών ζώων για την καλύτερη παραγωγή κρέατος. Ε, λοιπόν, ε, γίνεται ο ευνοχισμός, απαιτείται τέτοιου είδους παραγωγή από την άλλη θα, απαγόρευε, θα επιτρέψει την ελεύθερη βόσκηση, απαγορεύει τον ευνοχισμό κλπ. Ε, λοιπόν, μακρηγόρησα τώρα, ε, Ήμουν πιο σύντομος πριν, οπότε ζητώ λίγο την ανοχή σας που μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ. κυρία Ροντρίγες. Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν για τα κατάλοιπα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι μηδενικά τα κατάλοιπα στις βιολογικές εκμεταλλεύσεις. Έχουμε όμως και τις ε, παραγωγές, ε, τις καλλιέργειες με, ε, προϊό, με μεταλλαγμένους οργανισμούς. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να απαγορευτούν ολοσχερώς οι μεταλλαγμένες καλλιέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι αδύνατη, αδύνατος ο έλεγχος της επιμόλυνσης. Είναι αδύνατο να προστατεύσουμε πλήρως τις βιολογικές καλλιέργειες από τις συμβατικές. Οπότε φανταστείτε, αν έχουμε και μεταλλαγμένους οργανισμούς επιπλέον, θα χάσουμε τελείως τον έλεγχο. Επίσης, όπως σας είπα, την ευθύνη του ελέγχου τη φέρουν οι ίδιοι παραγωγοί, αδίκως κατά τη γνώμη μου. Μιλήσατε και για τις μικτές καλλιέργειες. Εγώ πίστευα αρχικά ότι θα πρέπει να είναι αμυγής οι καλλιέργειες, αμυγός βιολογικές δηλαδή. Στην Ισπανία όμως έχουμε για παράδειγμα πρόβατα που όταν βοσκούν βοσκούν σε χορτονομές, σε βοσκοτόπια που δεν είναι βιολογικά. Καλλιεργούν παρόλα αυτά κτηνιατρικά φυτά, ε, καλαμπόκι, σίτο. Οπότε έβαλα κάπως νερό στο κρασί μου σε ό,τι αφορά την απέτηση που είχα να είναι αμυγός βιολογική μία παραγωγή. Πάντως η συνύπαρξη, ο συνδυασμό βιολογικής και μη βιολογικής καλλιέργεια ίσως δημιουργήσει πρόσφορο έδαφο για απάτες. Τώρα, για τις ε, εξαγωγές. Ε, οι οριακέ τιμέ θα πρέπει να είναι αυστηρέ και κατηγορηματικές για να αποφύγουμε τα σκάνδαλα και τις απάτες. Θα πρέπει να ισχύουν για τα εισαγόμενα προϊόντα ίδιες υψηλέ και αυστηρέ προδιαγραφέ με τα ε, ενδοκινοτικά προϊόντα. Δεν ξέρω αν είναι εύκολος βέβαια ο έλεγχος, γιατί μιλάμε για μαζικές εισαγωγές. Δεν έχουμε λίγα κιλά εισαγόμενων προϊόντων. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε αναλυτικό έλεγχο όλων των εισαγόμενων προϊόντων. Άλλη ερώτηση για τους σπόρους. Είπα ότι στην Ισπανία είναι δύσκολο να αγοράσει ένας βιοκαλλιεργητής πιστοποιημένους σπόρους. Δεν έχουμε στην Ισπανία, προσφεύγουμε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα να αγοράσουμε αυστριακούς ή γερμανικούς σπόρους, αλλά δεν, προσαρμόζονται, δεν είναι προσαρμοσμένοι στις ε, γεωγραφικές ε, και εδαφολογικές ισπανικές ιδιαιτερότητες. Δεν ευδοκιμούν οι ίδιοι σπόροι παντού. Γι' αυτό θα πρέπει ο κανονισμός να διευκολύνει τους γεωργούς να παράγουν τους δικούς τους σπόρους χωρίς υπερβολική επιβάρυνση γραφειοκρατική. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ήταν ε, καταπληκτικές ε, όλες οι παρεμβάσεις. Μας τροφοδότησαν ε, με πολλές πληροφορίες και θα εμπλουτίσουν και τη δική μας συζήτηση και τις γνώσεις μας. Αν έχετε και άλλες ερωτήσεις μπορούμε γραπτώς να τις στείλουμε στους εμπειρογνώμονές μας και να μας στείλουν και αυτοί γραπτώς τις απαντήσεις τους. Ευχαριστώ και πάλι τους καλεσμένους εμπειρογνώμονες και να ξαναδώσω το λόγο για πολύ σύντομο διάστημα όμως ένα λεπτό στον εισηγητή μας τον κύριο Χόισλινγκ. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλου του συζητητέ αυτή τη ακρόαση, διότι πιστεύω πω ήταν πάρα πολύ σημαντικό να καλέσουμε εδώ εμπειρογνώμονε, έτσι ώστε να μα εκθέσουν ακριβώ πώ έχει η κατάσταση. Και πιστεύω πω η κριτική ήταν ενιαία. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεπεράσει τα όρια του αναγκαίου και πιστεύω πω όλοι εδώ συμφωνούμε ότι δεν θέλουμε μια ολική αναθεώρηση, αλλά μια περαιτέρω επεξεργασία και εξέλιξη του φυστάμενου κανονισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίγον να ε, υποδείξουμε στην Κομισιόν τις ε, επιθυμίες μας. Προτού έχουμε μία ε, πρόταση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον της οικολογικής αγεωργίας και το μέλλον αυτό χρειάζεται και έναν σωστό κατάλληλο κανονισμό. Αυτός ο κανονισμός δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με αυτή την μορφή της πρότασης και ελπίζω να ε, καταφέρουμε να κάνουμε ε, ολοκληρωμένες και σωστές ε, προτάσεις. Και θα ήθελα να πω ότι δεν είναι η Κομισιόν αυτή που επινόησε και ανακάλυψε την βιολογική γεωργία, αλλά είναι οι ίδιοι οι βιολογικοί αγρότες, οι καλλιεργητέ εκείνοι οι οποίοι πρωτοπορούν στον τομέα και εκείνοι είναι επίσης και οι αρμόδιοι για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωσή του. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω ξανά όλους εσάς που ήρθατε εδώ και ελπίζω να οδηγηθούμε όλοι σε, μια, σε έναν κοινό στόχο γιατί είναι προς το συμφέρον όλων μας. Ο τομέας έχουμε καταλάβει όλοι ότι χρειάζεται σαφέστατο πλαίσιο, σαφέστατες νομικές διατάξεις που θα τον βοηθούν και θα τον υποστηρίζουν παρά να τον εμποδίζουν. Σας ευχαριστούμε κύριε Χόισλινγκ. Ευχαριστούμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρακολούθησε τη δημόσια κρόαση και θα σημείωσε κατά λεπτός όλες τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Μία σύντομη διακοπή και σχεδόν αμέσως μετά θα περάσουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Παρακαλώ να εγκαταλείψετε γρήγορα και αθόρυβα την αίθουσα.